Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τώρα τη συνεδρίασή μας και με συγχωρείτε ζητώ συγγνώμη από τους Γερμανούς διερμηνείς θα μιλήσω αγγλικά από φιλοφρόνηση για τον τιμόμενο προσκαλεσμένο μας τον κύριο Φίλ Αγγελίδη ο οποίος είναι ο πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής Ερεύνησης Οικονομικής Κρίσης η οποία είχε καταρτιστεί τον Μάιο του 2009 και δημοσίευσε ε, τις 13 ε, Ματίου την ε, ε, έκθεσή του. Ε, είχαμε γνωρίσει τον κύριο Αγγελίδη όταν είχαμε πάει στη Washington για να συναντήσουμε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη. Είχαμε συναντηθεί τότε και ήδη είχαμε ανταλλάξει απόψεις. Βέβαια, εντωμεταξύ ο Φιλ τέλειωσε την εργασία του, παρουσίασαν τα πορίσματά τους και ε, εμείς τώρα ξεκινούμε να καταρτίζουμε την τελική μας έκθεση ε, κυκλοφορούν οι τροπολογίες και αύριο και σε μερικές εβδομάδες θα συζητήσουμε την πρόοδο της δικιάς μας εκθέσεως αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ο Φίλ Αγγελίδης είναι ε, ένας γνωστός μια γνωστή προσωπικότητα στις Ηνωμένε Πολιτείες με πολύ μεγάλη πείρα από πλευρά προστασίας ε, σε θέματα ε, οικονομικά ε, ήταν ο μίας ε, εις ε, την διοίκηση της Καλιφορνίας σε επίπεδο πολιτείας η οποία έχει ένα ε, τεράστιο, ένα τεράστιο αποθεματικό και έμεινε εκεί ως το 2007 και όπως σας είπα τώρα εδώ και 1,5 χρόνο ήταν πρόεδρος αυτής της Επιτροπής και έκτοτε ασχολήθηκε με οικοδομικά αφού έφυγε δηλαδή από τις δημόσιες υπηρεσίες. Του δίνω τον λόγο τώρα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ. Ε, uh, Πρόεδρε Κλίντς, ευχαριστώ, ευχαριστούμε που με καλέσατε να εμφανιστώ σήμερα ενώπιον της Επιτροπής σας και να συζητήσουμε αυτήν την τελική εκδοχή της εκθέσεως για την Ερωτική Επιτροπή. Και ε, ε, κατά αυτόν τον τρόπο δούμε τι έγινε και όσον αφορά αυτή τη ε, μεγαλύτερη κρίση που έχουμε γνωρίσει από τότε που είχαμε τη μεγάλη ύφεση. Ο σκοπό μα είναι να δούμε τι έγινε. Ε, είχατε έρθει τότε και στην Washington η Επιτροπή για την κρίση και αυτό είναι κομμάτι από τον συνεχιζόμενο διάλογο, το διαρκή, τον πάγιο διάλογο μεταξύ ημών και ημών, ώστε να δούμε αποτελεσματικά πώ θα προστατεύσουμε καλύτερα το χρηματοπιστωτικό μα σύστημα και την οικονομία μα. Επομένω, σήμερα να κάτσουμε και να δούμε πρώτα-πρώτα. Έχω μια εισήγηση και κατόπιν να συζητήσουμε ρωταπαντήσει και να κάνουμε ένα διάλογο να ερωτηθεί ό,τι θεωρείτε εσεί κύριε Πρόεδρε. Ο σκοπό τη δική μα Επιτροπή ήταν να ξεκαθαρίσουμε το τι έγινε και πώ συνέβη, ούτω ώστε να κατανοήσουμε γιατί συνέβη. Πιο συγκεκριμένα, μα ανέθεσαν ε, το, το, το Κογκρέσο, δηλαδή και ο πρόεδρό μα, να ε, ε, δούμε ποιε είναι οι αιτίε από αυτήν την χρηματοπιστωτική κρίση στι ΗΠΑ και επίση να διερευνήσουμε το γιατί είχαμε κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία ε, κατέρευσαν και επίσης γιατί κάποια άλλα αν δεν είχαν ενίσχυση και αρρωγή και και από την κυβέρνηση θα είχαν καταρρεύσει. Επίσης θα πρέπει να δούμε ε, ότι ε, μας ανέθεσαν να καταγγείλουμε στις δικαστικές και εισαγγελίες αρχές της χώρας μας ότι παραβάσεις του νόμου διαπιστώσαμε ότι έχουν ε, γίνει. Αυτά και κάναμε οπότε ε, παρουσιάσαμε στο Κογκρέσο τα συμπέρασματά μας στις 27 πρώτο φέτος. Κάναμε μια εξαντλητική ε, έρευνα και κράτησε αυτή η έρευνα πάνω από ένα χρόνο. Κατά αυτή μα την έρευνα ε, χρησιμοποίησαμε, διαβάσαμε εκατομμύρια σελίδων, εξετάσαμε 700 μάρτυρες και είχαμε επίσης δημόσιες ακροάσεις που εκράτησαν 19 μέρες. Οπότε είχαμε την δημοσίευση, εκτύπωση και σε ηλεκτρονική μορφή αυτή μα αυτής μας της και επίσης είχαμε χιλιάδες από έγγραφα. Είχαμε επίσης ε, τις καταθέσεις, είχαμε κασέτες, είχαμε αποτύπωση σχετική τέλο πάντων των καταθέσεων και, και, και άλλων συνεντεύξεων και όλα αυτά ε, μπορείτε να τα βρείτε ε, στο website το οποίο έχουμε να σας πω ποια είναι η ηλεκτρονική διάθεση του website που έχουμε Α, άλλαξε, άλλαξε Τώρα μόλις είναι το εξής fcic.lw.stanford.edu και επαναλαμβάνει ο μιλητής FCIC Law Stanford EDU και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιτροπής μας στις 13 Δευτέρου. Οπότε ε, προσπάθησαν λοιπόν να πούν κάποιοι ότι μπορούν να σβήσουν την μνήμα σε αυτό το οποίο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τι εξελίξει. Όμω, εγώ θεωρώ ότι αν δεν διδαχθούμε, ε, αν δεν αντλήσουμε συμπέρασμα την ιστορία, τότε δεν είναι δυνατόν ποτέ να μπορέσουμε να συγκροτηθούμε, να, να, να ορθοποδήσουμε και πάλι. Και στη συνέχεια, επομένω, αυτή τη κατεύθυνση προσπαθούμε εμεί να δούμε τα πραγματικά περιστατικά, τι ευθύνε, του μύθου, να καταλάβουμε πώ θα αποφεύγουμε την ε, κρίση αυτή. Και προσπαθούμε, επομένω, όχι να ξαναγράψουμε την ιστορία, άρα να την καταγράψουμε. Και ούτε θέλουμε όμω κανεί να την ε, παραχαράξει την ιστορία, τα πράγματα δύο όπω έγιναν. Είχαμε αυτή την παγκόσμια κρίση επομένω, η οποία φυσικά έχει σοβαρέ συνέπειε και για τη ΣΥΠΑ και για τι χώρε όλε παγκοσμίω. Όλοι επομένω περιμένουμε πώ και πώ να υπάρξει ανάκαμψη, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι είχαμε ε, αυτού του είδου του κλειδονισμού τη οικονομία και οι οποίοι χτυπήσαν μια ολόκληρη γενιά. Διότι χτύπησαν τι επιχειρήσει, ε, κοινότητε, νοικοκυριά και εδώ και στην Ευρώπη και στη χώρα μα, επομένω και στην Ευρώπη. Οπότε εμεί ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από του μετασυσμού ε, αυτή τη καταστροφή και είχαμε πάνω από 26 εκατομμύρια Αμερικάνου οι οποίοι χάσαν τη δουλειά του ή που δεν μπορούσαν να βρουν πλήρη απασχόληση ή που παρετήθηκαν από το να ψάχνουν για δουλειά. Είχαμε περίπου 11-3 όσον αφορά τις ε, αποταμιεύσεις οι οποίες χάθηκαν. 4 εκατομμύρια ήταν οι οικογένειες που ε, χάσαν τα σπίτια τους τα οποία κατεσχέθησαν λόγω της ε, κρίσης και επίσης λένε ότι θα πάμε για τα 8 έως 13 εκατομμύρια οικογενειών που θα υποστούν το ίδιο. Επίση, έχουμε διάφορου αθώου, κάποιοι δηλαδή οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα παράνομο, τίποτα κακό, οι οποίοι τώρα τρέμουν για το μέλλον και νιώθουν πλήρη ανασφάλεια. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ε, συζητούμε συνέχεια κατάπαστα για το, αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση. Δηλαδή το να προσφέρει ένα δεκανίκι ενίσχυση αρρωγή σε χρηματοπιστικά ιδρύματα τα οποία θεωρήθηκε ότι είναι τόσο σημαντικά, τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να καταρρεύσουν. Όμω αυτό το οποίο ήταν δική μα αποστολή είναι να εξετάσουμε ε, μια, ένα, θέμα πάρα βασικό. Το 2008 τι έγινε, γιατί έπρεπε να διαλέξουμε μεταξύ ε, δύο πάρα πολύ σκληρών εναλλακτικών λύσεων. Μεταξύ σκύλα και χάρη είμαστε. Δηλαδή έπρεπε να καταρρεύσει η οικονομία και οι ή θα έπρεπε να ρίξουμε τρισεκατομμύρια από δολάρια των φορολογούμενων στο σύστημα και στι ε, ιδιωτικέ εταιρείε, παρά το ότι ε, είχαμε εκατομμύρια που χάναν τη δουλειά του, χάναν τι αποταμίε του, χάναν τα σπίτια του. Και τελικά φτάσαμε στα εξή έξι συμπεράσματα και θα σα πω με δύο λόγια ε, αυτά τα, τα έξι σημεία στα οποία καταλήξαμε. Πρώτα-πρώτα, συμπέρασμά μα ήταν ότι θα μπορούσε να αποφευθεί αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση παρά τα όσα είπαν πάρα πολλοί στου ε, χρηματοπιστωτικού και πολιτικού κύκλου ότι δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί η κρίση. Υπήρχαν πάρα πολλά σημάδια τα οποία προδοποιούσαν. Επομένω, ε, το ότι η τραγωδία είναι ότι, ότι κανεί δεν τα υπολόγισε, ε, δεν τα έλαβαν υπόψη, τα, τα και επομένως εμείς το είπαμε αυτό κατηγορηματικά. Ούτε, ούτε, ούτε, καν κομπιούτερ τρελάθηκε, ούτε φταίει η φύση, ούτε είχαμε καμιά αρχαιομηνία. Επρόκειτο για αυτού που κρατούσαν τα ενία τη οικονομία, επρόκειτο για του για τους πολιτική της πολιτικής τη ζωής, ζωή, ζωής, οι οποίοι αγνόησαν αυτά τα σημάδια και έτσι ε, φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση που τόσο έμπλεξε την, την ευημερία μας. Επομένως, δεν ε, πρόκειτο για, για, για, για κάποιον που σκόνταψε, ε, πρόκειτο για κάποιον που το τα πήγε τελείως λάθος. Είχαμε επομένω τα subprimes αυτά, τα οποία ξεκίνησε το, τη διαδρομή τους τα τέλη του, της δεκαετίας του 90 και είχαμε διάφορα, διάφορα δάνεια τα οποία ήταν καταπλεονεστικά και το 2004 το FBI είχε πει ότι ενδημούσε φαινόμενο ε, στεγαστικών δανείων τα οποία όμως είχαν πάρα πολύ ε, όρου. όρους και επομένως έλεγαν ότι θα οδηγηθούμε σε αυτή την κρίση τέλος ε, της δεκαετίας του 80 και αρχής της δεκαετίας του 90 και άλλα σημάδια υπήρχαν δηλαδή ε, είχαμε τα παράγωγα εξε, εξεράγει αγορά κάποιο τρόπο το ίδιο έγινε επίσης και με την ε, εμπιστοσύνη των των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ε, αυτό ε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος και κανείς δεν έκανε τίποτα ούτω ώστε να φρενάρει αυτή την πορεία προς την χρηματοπιστωτική κρίση. Έχουμε ένα σωρό αποτυχίες, ένα σωρό λάθη, διότι πρώτα-πρώτα η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, το Federal Reserve, δεν έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουν σαν αυτά τα τοξικά στιγαστικά δάνεια. Επίσης, οι τράπεζες και τα συναφή ιδρύματα αγόρασαν διάφορα χαρτοφυλάκια για, χωρίς να εξετάσουν πόσο επικίνδυνα ήταν. Αυτό ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2006 και ε, πήγαμε στο, στη, στο 1,63 δολάρια τα οποία διατέθησαν ακριβώς σε τέτοια δηλητηριώδη δάνεια από το 2007 οι Moody's είχαν πει ε, ότι 45.000 ε, ε, χρηματιστηριακοί τίτλοι ήταν αλφα-αλφα-αλφα. Ε, και αυτό έγινε μέχρι το 2010 φτάσαμε να έχουμε τέτοιους αξιολόγους μόνο το 2006 η Μούντις ενέκρινε ένα σωρό τέτοια, ε, τέτοιους τίτλους τα τραγικά ήταν τα αποτελέσματα επομένως ποιο θα είναι το μεγαλύτερο λάθο σήμερα να πει κανένα ότι πρόκειται για κάτι αναπόφευκτο και ότι τίποτα δεν μπορούσε να κάνει κανεί Εάν πούμε ναι σε μια τέτοια σκέψη, τότε θα ξαναπάθουμε τα ίδια. Δεύτερο συμπέρασμα. Είπαμε ότι όλες, όλα αυτά τα λάθη όσον αφορά την ε, νομοθεσία, όσον αφορά την εποπτεία, ήταν τραγικά όσον αφορά ε, τι ε, αγορέ μα την οικονομία μας. Είναι σαφές ότι αυτοί που πρέπει να προσέχουν δεν προσέχανε. Αυτό ε, έγινε γιατί όλοι πιστεύανε κράτοντα ότι υπάρχει αυτορύθμιση στις αγορές και ότι υπάρχει κάποιο είδους ε, εποπτεία από τα ίδια τα χρηματοπιστικά ιδρύματα. Όμως ε, ο Greenspan αυτό πίστευε και εκείνος ο πρόεδρος της διοικητής δίκης μας τράπεζας αλλά και άλλοι, και άλλοι στο Κογκρέσο. Εμείς λέμε ότι εδώ πέρα υπήρχαν κάποια πάρα πολύ μεγάλα κενά όσον αφορά το σύστημά μας τότε, το τυθωράκι του συστήματος, γιατί είχαν τεθεί σε κίνδυνο 3 εκατομμύρια δολάρια. Ε, είπαμε, ήταν, επρόκειτο για τα παράγωγα και είπαμε για ένα σωρό μηχανισμούς που τελικά απαιτέλεσαν αυτό που λέμε σκιώδες τραπεζικό σύστημα, μαύρο τραπεζικό σύστημα. Επίσης και άλλες ε, ε και άλλα λάθη από πλευρά ομοσπονδιακών αρχών που δεν ε, ίσκησαν την εποπτεία που έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, δεν δεχόμαστε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ακόμα και με αυτές τις ελλείψεις και τα κενά είχαν αρμοδιότητες, είχαν εξουσία, αλλά επέλεξαν να μην την ασκήσουν, να μην τη χρησιμοποιήσουν τι αρμοδιότητες τους και θα έπρεπε επομένω και όπου δεν είχαν τις αρμοδιότητες να, να φροντίσουν να τις αποκτήσουν για να ασκήσουν την εποπτεία που έπρεπε. να σας πω τώρα ε, πώς θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα ήταν η μόνη που μπορούσε να σταματήσει αυτού του είδους το, το, το, ξέφρενο δανεισμό θα έπρεπε να μπορούν, ε, μάλλον μπορούσαν, μπορούσαν, είχαν τις πληροφορίες και μπορούσαν επομένως να ε, βγουν μπροστά και να σταματήσουν το φαινόμενο. Δεν το κάναν όμως. Επίσης, η Χρηματιστηριακή Επιτροπή, Securities και Exchange Commission, επίσης μπορούσε να κάνει κάτι και δεν το έκανε. Ε, η Τράπεζα της Νέας Υόρκης και άλλες ρυθμιστικές αρχές επίσης μπορούσαν κάτι να κάνουν και δεν το έκαναν επίσης οι, αυτοί, οι ρυθμιστικές αρχές, η, η κυβέρνηση μπορούσε επίσης ε, να σταματήσει αυτού του είδους τα στεγαστικά καταπλεονιστικά δάνεια γιατί υπήρχαν όλα τα σημάδια ότι πρέπει να το κάνουν και δεν το κάνανε. Ε, οπότε βλέπουμε ότι συνέχιζαν να αξιολογούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ω υγιή ενώ δεν ήταν, ενώ υπήρχαν όλε οι ενδείξει περί του αντιθέτου. Να πώ έγινε η κατάρρευση αυτών. Λοιπόν, ε, γι' αυτό και δεν μα ε, εξέπληξε το ότι η, αγορά συνέχεια ήθελε όλο και λιγότερη ρύθμιση. Όμω κανένα δεν, δεν παρενέβη, κανένα δεν, δεν εφήρμοσε του νόμου και έτσι επομένω το κράτος μας δεν είχε την, την εποπτεία που θα απαιτούσε ένας τόσο σημαντικός κλάδος, η οικονομία. Και τελικά οι, οι ηγέτες μας ε, ουσιαστικά μας πρόδωσαν. Τρίτον, διαπίστωση η Επιτροπή μας ότι όλες αυτές οι τραγικές ε, αποτυχίες ε, όσον αφορά την διακυβέρνηση και τη διαχείριση ήταν το κλειδί, ήταν η απάντηση, ήταν η εξή γιατί έγινε η κρίση. Είχαμε απορρίθμιση που κράτησε 30 χρόνια. Είχαμε το χρηματοδοτικό σύστημα το οποίο έτσι είχε ε, αδυνατήσει ε, και αυτό είχε επίδραση στον τρόπο του επιχειρήν από τους πάντες στην αγορά. Και επίσης είχαμε κάποιες εταιρείες οι οποίες θεωρούσαν ότι ε, ότι, ότι, και θεωρήθηκε μάλλον ότι αυτές οι εταιρείε από μόνες τους θα, θα επόπτευαν τον, τον εαυτό τους. Όμως εμείς είδαμε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα και είχαμε πάρα πολύ μεγάλα λάθη ε, τα οποία φάνηκαν στο τι με την AIG, την ε, Bear Stearns, την, την Fannie Mae, Lehman Brothers, Mary Lynch και άλλους πολλούς. Οπότε φτάσαμε σε κάποια φιλοσοφία, σε κάποιες αποφάσεις πάρα πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολλές από αυτές τις ε, εταιρείε ε, ενήργησαν με, πάρα πολύ, ε, με βαρέως αμήλη τρόπο γιατί πήραν μεγάλα ρίσκα, διέθεταν λίγο κεφάλαιο και εξαρτήθηκαν πάρα πάρα πολύ από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Τελικά, βλέπουμε ότι έγιναν κάποιες αλλαγές στις τράπεζες, στις επενδυτικές, στους όμιλους εταιριών και πρόκειται για τις εταιρείε οι οποίες εκτέθηκαν πάρα πολύ όσον αφορά τα subprimes και όσον αφορά ε, τι, τις, ε, τις συναλλαγές σε χρηματιστηριακούς τίτλους ε, που φτάνανε σε τάξη μεγέθους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε ανοιγόντουσαν συνέχεια, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το άνοιγμα. Και τελικά τι κάνανε. Αγνόησαν ακόμα και τα μαθηματικά μοντέλα όσον αφορά ε, την πρόβλεψη του κινδύνου. Επίσης, τα, στα αντισταθμιστικά συστήματα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ε, διακρινόντουσαν από ανταγωνισμό, ε, λίγη ρύθμιση, ισχυρή νομοθετική ρύθμιση και όλοι κοιτάγανε μόνο το, τις πιθανότητες κέρδους και όχι τις πιθανότητες του κινδύνου. Επίσης, τέθηκε τελείως εκτός ελέγχου το επιχειρήν με αυτά τα παράγωγα. Φτάσαμε στα 673 τρισεκατομμύρια το 2008. Ε, είχαμε επίσης ε, τα παράγωγα τα οποία ε, περνάγαν από το χρηματιστήριο, τα οποία και αυτά οδήγησαν στην κρίση. Ε, είχαμε τιμόχλευση, είχαμε έλλειψη διαφάνειας, είχαμε ε, πάρα πολύ λίγη εποπτεία όσον αφορά την επάρκεια κεφαλαίων οπότε ε, έτσι φτάσαμε σε μια φούσκα η οποία έσκασε, η οποία έσπασε και αφορούσε επίσης και τον κλάδο των κατασκευών μετά από αυτή την, την ε, κατάρρευση τελικά ήταν στην καρδιά της κρίσης τα, τα παράγωγα τώρα άλλο συμπέρασμα είναι αυτό το οποίο είπαμε το ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη ε, διακυβέρνηση, ούτε κατάλληλη νομοθεσία. Μέχρι το 2008 είχαμε πάρα πολλά δάνεια που είχαν πάρει οι τράπεζες. Δεν είχαν ε, επαρκή κεφάλαια, δεν είχαν επαρκή ρευστότητα. Οι βασικές μενικές τράπεζες, Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch και Morgan Stanley, είχαν πάρα, πάρα πολύ ε, ισχνή επάρκεια κεφαλαίων. Το 2007 η αναλογία της μόχλευσης ήταν 40 προς 1, τρομερό. Και σήμερα τη Γαλλία, όσον αφορά στοιχεία ενεργητικού, είχαν μόνο ένα δολάριο για να καλύψουν δεχόμενες ζημίες. Ακόμα χειρότερα. Η δανειοδότηση ήταν βραχυπρόθεσμη και γινόταν στην αγορά overnight. Άρα θα έπρεπε να δανείζονται κάθε μέρα, καθημερινά. Φάνη Μέη και οι άλλες είχαν, το, είχαν μόχλευση 75 προς 1. Η Citigroup 48 προς 1 το 2007. Αυτή η μόχρευση για τις τράπεζες πολλές φορές ε, κρυβότανε και για τα παράγωγα και με τις ε, εκθέσεις και σολογισμούς που δημοσιευόντουσαν. Τίποτα δεν λέγανε Έχουμε καταγραφή τέτοιων περιστατικών στην εκθεσή μας που αφορά και τη Lehman Brothers και την Bear Stearns και αυτοί απέκρουν την πραγματική κατάσταση. Επίσης, ακόμα και αν η αγορά των στερεωστικών δανείων όλο και περισσότερο, ε, σε περισσότερο κίνδυνο βρισκόταν, οι εταιρείε και οι τράπεζε αυτέ συνεχίζανε να προχωράνε τον ίδιο τρόπο. Όμω δεν ήταν μόνο οι τράπεζε. Και τα νοικοκυριά κάνανε το ίδιο. Επομένω, ήταν ολοένα και μεγαλύτερε πιθανότητε το σύστημα να καταρρεύσει. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου προστασία Ακριβώς όπως έγινε στην αρχή του 20ου αιώνα. Να υπάρχουν κάποιο είδους φράγματα σε μια τέτοια πλημμυρίδα του φαινομένου, δηλαδή της κατάρρευσης. Μιλάμε για ε, πρόβληματα της τάξης των 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν υπήρχε επομένως διαφάνεια. Υπήρχαν μεγάλα χρέη τα οποία σωρεύθηκαν, ανεπάρκεια κεφαλαίου και στοιχεία ενεργητικού τα οποία ήταν πάρα πολύ επισφαλή. Επομένως ακολούθησε ο πανικός και θερήσαμε τις θέλες πως πήραμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι λοιπόν, για την κρίση. Ούτε μπορέσαμε να βρούμε τις απαντήσεις όταν αυτή ξέσπασε. Ο Υπουργό Πόλσον, ο Άλαν Γκρίνσπαν και κατόπιν ο Μπερνάγκη στην Κεντρική Τράπεζα και ο Τιμ Γκάτνερ από πλευρά τη ε, Reserve Bank τη Νέα Υόρκη εξεπλάγησαν. 2007 και 2008. Και ήταν τα χέρια τους διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γινόταν με το σύστημα το οποίο διαχειριζόντουσαν. Επομένως, επρόκειτο περί αμέλειας και έλλειψης διαφάνειας. Θεωρούσαν ότι είχαν κατανομή των κινδύνων, ενώ συνέβαινε το αντίθετο. εκεί δεν είχαν συγκεντρωθεί στο ίδιο σημείο. Και όσο περισσότερο τα subprimes απειλούσαν το σύστημα, προσπαθούσαν με το λάθος τρόπο να ανασχέσουν τον κίνδυνο. Δεν υπήρχε ένα γενικό σφαιρικό στρατηγικό πλάνο. Και έτσι χτυπήθηκαν οι... Και έτσι χτυπήθηκε η χρηματοπιστωτική αγορά. Επίσης είπαμε ότι η φούσκα των ακινήτων απειλούσε όλο το σύστημα. Παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2007 τα hedge funds της Bear Stearns αυτά τα οποία είχαν ε, συνδεθεί με στεγαστικά δάνεια κατέρευσαν. Θεωρήθηκε ότι αυτό ήταν απομονωμένο φαινόμενο. Άλλο παράδειγμα, η Federal Reserve της Νέας Υόρκης ακόμα έψαχνε ενημέρωση για το πόσο είχε εκτεθεί η Lehman Brothers μόλις ένα μήνα πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers ενώ υπήρχαν στο παιχνίδι 900.000 παράγωγα. Αποφάσισε η κυβέρνηση να διασώσει την Bear Stearns και τότε έβαλε τη Fannie Mae και τον Freddie May, τη Fannie Mae σε επιτήρηση, ε, και ακολούθησε γρήγορα η αποφάσιση να, απόφαση να αφήσουν να καταρρεύσει η Lehman. Και αυτό οδήγησε σε πανικό στην αγορά και αμβεβαιότητα. Και έκτον και τελικόν η έκθεσή μας εξηγεί πώς παραβιάσουν αφορά την διοντολογία και τον έλεγχο ε, διαδέθησαν σε όλα τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της ε, πρώτης κρίσεως. Η ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών μας αγορών και τη πίστεω του κοινού σε αυτέ τι αγορέ είναι πολύ βασικά στοιχεία για την ευμάρεια. Η ευμάρεια του χρηματοστικού συστήματο και τη οικονομία μα βασίζονται σε έννοιε όπω είναι οι δίκαιε συναλλαγέ, η ευθύνη και η διαφάνεια. Εκεί βασίζεται και ορθότητα τη λειτουργία του συστήματο. Μετά από προσεκτική έρευνα και ε, διαπιστώσαμε ότι αυτή η κρίση τροφοδοτήθηκε από συστημική κατάρρευση όσον αφορά τη δοντολογικό κανόνα που εφαρμοζόταν ε, και ε, σε όλα τα επίπεδα μέχρι τα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων χρηματοστικών εταιριών. Λοιπόν, αυτό κατέληξε όχι σημαντικέ χρηματοστικέ συνέπειε, αλλά επίση σε απώλεια εμπιστοσύνη από πλευρά επενδυτών επιχειρήσεων και του κοινού. Παραδείγματα αυτών των παραβιάσεων συμπεριλαμβάνουν ότι οι δανειστέ οι οποίοι δεν πλήρωσαν τα στεγαστικά του δάνεια και τόσο γρήγορα αφού πήραν το δάνειό του, και αυτό έδειχνε ότι ποτέ δεν είχαν τη δυνατότητα ή την πρόθεση να πληρώσουν τα στεγαστικά του δάνεια. Οι μεσολαβητές όσον αφορά ε, τους, ε, τα στεγαστικά δάνεια. Ε, συνεργάστηκα με τους δανειοδότες και με τους δανειοδότες σε, ψηλό, σε δάνεια ψηλού κόστους ώστε να πάρουν μεγάλα τέλη. Λοιπόν, άνθησε η απάτη στον τομέα αυτών, διότι δεν, ήταν, δεν εφαρμόστηκαν οι προδιαγραφές και οι νόμοι. Μια μελέτη έδειξε ότι ήταν πάνω από ένα τρισεκατομμύρια δολάρια δανείων στεγαστικών που στα πλαίσια απατών που δόθηκαν μεταξύ 2005 και 2007 και το αποτέλεσμα ήταν απώλειες πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εταιρείε όπως η Goldman Sachs δημιούργησαν και πώλησαν ε, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια τίτλους ε, ως ασφαλίσεις όσον αφορά στεγαστικά δάνεια στους επενδυτές. Και τελικά, όταν τελικά οι χρηματοστικές εταιρείε πολλούσαν αυτούς τους, ε, αυτές τις δανειοδοτήσεις με ψηλό κίνδυνο, ε, δεν έδιναν πληροφορίες όσον αφορά την ποιότητα των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται. Θα ήθελα να πω ότι αξιολογώντας ε, τις ευθύνες είδαμε ότι οι δημόσιοι ηγέτες που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των φυσικών συστημάτων ήταν βασικά υπεύθυνοι. Αυτοί που έπρεπε να διευθύνουν τους ρυθμιστικούς φορείς και οι διευθυντές των διαφόρων εταιριών που θα μπορούσαν να λέξουν την κρίση. Ο νόμος δεν μας ανέθεσε να κάνουμε συστάσεις όπως η Επιτροπή Κρίς, αλλά ο σκοπός της εκθέσεώς μας ήταν να αποτιμήσουμε τα όσα συνέβησαν, ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε νέα ρότα. Ε, καταστήσαμε σαφές ότι η έκθεσή μας δεν θα πρέπει να ειδωθεί στο τον τέλος ε, των ερευνών για την κρίση που γίνονται στη χώρα μας. Πάρα πολλά μπορούμε να μάθουμε, πολλά να ερευνήσουμε, πολλά να διορθώσουμε και από πολλές τυχές το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα που έχουμε σήμερα εξακολουθεί να είναι μετάβλητο αν συγκρίσει με αυτό που υπήρχε τις παραμονές της κρίσης. Και πράγματι υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού και λιγότερη χρηματοστατικά ιδρύματα συστημικά σημαντικά από πριν. Σύμφωνα με τον φορέα τη Νέα Υόρκη, τα κέρδη του χρηματοδοτικού τομέα με το τέλο του 2009 έφτασαν τριπλάσια επίπεδα του 2006 και η επίπεδα αποζημιώσεως για δημόσιες, ε, δημόσιες ανταλλαγές τίτλων έφτασαν νέα ρεκόρ το 2010. Πριν ε, ολοκληρώσω την παρέμβαση σήμερα, θα ήθελα να εκφράσω κάποιε προσωπικέ παρατηρήσει πέραν από αυτέ που συμπεριλαμβάνονται στην εκκλησία μα όσον αφορά ποια είναι η χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στη χρηματοστική αγορά δύο μήνες μετά την έκθεσή μας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των ερευνών μας διαπιστώσαμε ότι πολύ λίγη αυτοκριτική ασκήστηκε από την Wall Street όσον αφορά τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν και το ρόλο που η Wall Street αυτό οφείλεται κατά πολύ στο ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι έτρεξαν στη διάσωση του χρηματοδοτικού ε, συστήματος και διάφορων χρηματοδοτικών επιχειρήσεων και έδωσαν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω περίπου 24 προγραμμάτων οικονομικής αρρωγής της κυβερνήσεως. Και έτσι η Wall Street σε μεγάλο βαθμό δεν χρειάστηκε να υποστεί τις συνέπειες των σφαλμάτων της και επανεξέταση που θα έπρεπε να κάνει πληρώνοντας τις συνέπειες. Ε, πολύ δημόσια προσοχή εστιάστηκε επί των 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκαν στο πρόγραμμα του STARP. Αυτό το πρόγραμμα πολλέ πτυχέ ήταν η κορυφή του παγόβουνου ενό άνευ προηγουμένου αποτολμήματο τη ε, κυβερνήσεω να διασώσει το χρηματοστικό τομέα από κατάρρευση. Και πιο σημαντικά φαίνεται να μην υπάρχει σχετισμό μεταξύ εκείνων που οδήγησαν τη χώρα μα και τον κόσμο στην οικονομική κρίση με εκείνου που πληρώνουν τελικά για την καταστροφή με πολύ λιγέ ή ελάχιστε μηδενικέ συνέπειε για εκείνου που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την θύελα αυτή που περνάμε. Σε αυτά τα πλαίσια, οι παρούσε προσπάθειες που έχουν δρομολογηθεί από τον εκδοτικό τομέα και τους πολιτικούς μα συμμάχου στις χώρες μας και στις προστεύουσες των ε, χωρών μα για να εφαρμόσουν ε, τις διάφορες προσπάθειε προσπάθειες ε, είναι ανησυχητικές. Ήδη στις τελευταίους μήνες είδαμε συγκεντρωμένε προσπάθειες να γυρίσουν πίσω το χρόνο των διαφόρων χρηματοστοικών ε, μεταρρυθμίσεων ε, ένα νόμο που έχουμε θεσπίσει που θα μας βοηθούσε να αποφύγουμε την ακρίση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων προσπάθησε να περικόψει τον προπολογισμό για τις επιτροπές για, τα, για τις μετοχές στον προσωπικό τομέα παρά το γεγονός ότι φορέας αυτός ε, μαζεύει περισσότερα από ό,τι προβλέπει προπολογισμό από τα διάφορα πρόστιμα που επιβάλλονται. Και γίνονται δραματικές περικοπές ε, όσον αφορά την Επιτροπή για τη Συναλλαγή Μετοχών που έχει το Ηράκλειο ναχθο. Ε, τελικά να ελέγξει την αγορά των παραγόγων, ε, να τη φέρει στη διαφάνεια και είναι μια αγορά που ξύστησε σε εκατομμύρια δολάρια. Ο Alan Greenspan, του τελευταίου μήνε, που ο οποίο έχει τι μεγαλύτερε ευθύνε όσον αφορά το να ηγηθεί, μάλλον αυτό ευθύνεται για την οικονομική καταστροφή σε μεγάλο βαθμό, ε, λέει ότι οι νέε ρυθμίσει που θεσπίζονται είναι σε φρενήρι ρυθμό. Και λέει και παραθέτει οτιδήποτε είναι ρυθμιστικό και ζητά να επιστρέψει στι παλιέ καλέ μέρε Τη ε, της, μια της κάθε κινδύνου είναι αυτό που γονάτισε το σύστημα. Η πολιτική του ήταν η ασφαλμένη συνταγή πριν από την κρίση και εξακολουθεί να είναι η σίγουρη συνταγή τώρα δοθέντως ότι τα στοιχεία τα συντριπτικά που έχουμε μαζέψει εμείς ε, δείχνουν ότι οι πολιτικές το οδήγησαν σε τέτοια μεγάλα σφάλματα και βλάβη. Αυτέ οι αντιδραστικέ δυνάμει μαζί με την νομισματική ισχύ του χρηματοστικού τομέα δεν πρέπει να υπερισχύσουν. Θα πρέπει να ανανεώσουμε τη δέσμευση να μεταρρυθμίσουμε τον τομέα αν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία η οποία να είναι υγιής και ισχυρή. Σχετικά με αυτό έχω τρεις σκέψει που μπορούν ίσω να σα οδηγήσουν κάποιε σκέψει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να επιταχύνουμε το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και να ενισχύσουμε την αποφασιστικότητά μα, ούτω ώστε οι ρυθμιστικέ και οι πολιτικέ αλλαγέ θα πρέπει να λάβουν χώρα. Ο νέο νόμο που πέρασε από το Κογκρέσο και υπεγράφει από τον πρόεδρο Ομπάμα θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρω. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα απαιτηθεί οι ρυθμιστικοί φορεί να έχουν επαρκεί πόρου, να έχουν δύναμη και πολιτική βούληση και ένα Κογκρέσο το οποίο εξασφαλίζει ότι κάνει τη δουλειά του, ότι κάνει δουλειά του και να μην προσπαθεί να σταματήσει. Επίση θα απαιτηθεί συνεχή επαγρύπνηση και προσαρμογή από όλου μα. Ε, προωθήσει τη ταχύτατα μεταβαλλόμενου φύσεω του κοινοτιστικού τομέα και θα απαιτηθεί η ισχυρότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ τη χώρα μα, τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και άλλων χωρών, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα ταιριάζει πολύ καλά σε μια παγκοσμιοποιημένη χρηματοστική βιομηχανία που δεν θα επιτρέπει το πλαίσιο αυτό, ο χρηματοδοτικό τομέα, να πιέζει μια χώρα η ομάδα χωρών και να βάζει τη μια χώρα εναντίον τη άλλη ει βάρο του γενικότερου δημοσίου συμφέροντο. Δεύτερη σκέψη που έχω να κράσω. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χρηματοδοτικοί μα νόμοι θα εφαρμόζονται δίκαια αλλά αναμφιβισβήτητα. Ε, η Επιτροπή μα δεν δημιουργήθηκε σαν κάποιο εισαγγελέα, αν θέλετε. Αλλά το ερώτημα που τίθεται συχνά σε μένα μετά από την θητεία μου που ήμουν πρόεδρος είναι πού είναι οι διώξεις γιατί κανείς δεν πλήρωσε το τίμημα εν ώψη όλων των οικονομικών ζημιών που συνέβησαν υπάρχει πάρα πολλή οργή οργή και ζητούν υπεύθυνα να τιμωρηθούν. Αλλά ο θυμό δεν είναι μια συνταγή για τη διαμόρφωση πολιτική. Δεν θα πρέπει να ζητάμε εκδίκηση, αλλά θα πρέπει να δεσμευτούμε να επιδιώκουμε την εφαρμογή της ευθύ, της, του νόμου, το ώστε το κράτος δικαίου να μην εξαιρεί κανέναν, ούτε και αυτού που είναι πλούσιοι και έχουν ισχύ. Οπότε αυτό να είναι κάτι το οποίο αποτρέπει αυτούς να κάνουν τα ίδια στο μέλλον. Επειδή το χρηματοδοτικό του σύστημα είναι παγκοσμία μελία, θα πρέπει από σκηνού να συνεργαστούμε, ώστε οι νόμοι να μην παραβιάζονται. Εάν παραβιαστούν, εκείνους που παραβίασαν, να τιμωρηθούν, ακόμα και σε συνοριακό επίπεδο. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να δεσμευτούμε να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμη οικονομία, όπου ο χρηματοστικός τομέας θα, θα συμμετάσχει σε αύξηση και ανάπτυξη. Το κεφάλαιο τίθεται τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης επιχειρήσεων και για τη δημιουργία ευμάρειας. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα νέο συνέστημα εταιρική ευθύνη, που θα χαρακτηρίζεται από δεντολογικό κώδικα που εφαρμόζεται. Η μεγαλύτερη τραγωδία τη τελευταία δεκαετία ποια είναι. Του πάρα πολλά χρήματα. Θέλαμε να δημιουργήσουμε τις εκατομμύρια δολαρίων σε τίτλους στεγαστικούς που δεν λειτουργούσαν σωστά, παρά να δημιουργήσουμε υποδομέ, τεχνολογία, καθαρή ενέργεια, που αυτά θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητά μα και τον πλούτο μα και να ενισχύσουν τι κοινωνίε μα. Τα χρόνια πριν από την κρίση, η οικονομία μα αφορούσε περισσότερο γέννηση χρήματο από το χρήμα, παρά το χρήμα να δημιουργεί αξία. Και παρά το ότι δεν παραβιάστηκε κάποιο νόμοι, οι δεντολογικοί κανόνε επιδεινώθηκαν με τρόπου που διάβρωσαν ίδια τη βάση της οικονομικής πρόοδου. Στις ΗΠΑ το, το ποσοστό των κερδών του χρηματοστικού τομέα ανέβηκε από το 15% το 1980 σε πάνω από 30% τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτό μέχρι το 2007 το ποσό του χρέους που εκρατείτο από το χρηματιστικό τομέα των ΗΠΑ πήγε από τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια στα 36 δισεκατομμύρια δολάρια δι, διπλασιαζόταν στο μερίδιο όσον αφορά το ποσοστό του σε σχέση με το ΑΕΠ. Από πολλές γίναμε μια χώρα που βασιζόταν στα μεγάλα στοιχήματα και δεν στοιχημάτιζε στην αξία. Είναι και, η ώρα να κάνουμε ξανά προσπάθειες, η οικονομία μας να έχει άλλους στόχους. Ο χρηματοδοτικός τομέας δεν θα πρέπει να είναι το αφεντικό, αλλά ο υπηρέτης της οικονομικής μας πρόοδου. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλη η θεωρία της κρίσης οικονομικής και χρηματοδοτικής που έπληξε τις χώρες μας ε, δεν έχει τελειώσει από κοινού θα έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε το τελικό κεφάλαιο και τώρα σε εμά εναπόκειται να κάνουμε διαφορετικέ επιλογέ αν θέλουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έρθω εδώ και να μιλήσω μπροστά σα. Uh, Ευχαριστώ, Φιλ, για αυτή την λεπτομερή εισαγωγή ε, στην έκθεσή σου και στα πορίσματα της εκθέσεώς σου διότι ουσιαστικά ήσασταν μια εξεταστική επιτροπή για την οικονομική κρίση, πράγμα που δεν είμαστε εμείς και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μας. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ της δικιάς σας και της δικής μας επιτροπής. Επίσης, ε, επιλέξαμε επιλέξατε στην Επιτροπή σας εξοκοινοβουλευτικούς συμμετέχοντες ενώ τα δικά μας μέλη είναι ευρωβουλευτές. Θα ήθελα λοιπόν τώρα καταρχήν να ζητήσω από τους εξπροσώπους των πολιτικών ομάδων να κάνουν ερωτήματα ή να κάνουν σχόλια και θέλω να ξεκινήσω πρώτα με το ΕΛΚ, μετά τους σοσιαλιστές σε δύο. Εσείς θέλετε να μιλήσετε πρώτα, βεβαίως. Πρώτα, πρώτα ε, η συγγήτρια, μετά δύο συντηρητικοί, δύο σοσιαλιστές, δεν βλέπω κανέναν φιλελεύθερο, έναν εκπρόσωπο της αριστεράς και από την ε, EFD και υπερβόνς όμως έχει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγγελίδη, παρακαλώ μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά σας, διότι θα μιλήσω γαλλικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ μετά την επίσκεψη που είχαμε κάνει εις την Αμερική και ε, στην εργασία η οποία περιμένει, ε, μας περιμένει ακόμη είναι πολύ βασικά τα πορίσματά σας γι' αυτό θα κρατήσω μόνο δύο από αυτά προσχόλιο καταρχήν ότι πολλούς από αυτούς που φέρουν μεγάλη ευθύνη είναι αυτοί οι οποίοι τώρα είναι υπεύθυνοι για να βρουν και τις λύσεις πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα αλλάξουν και πολλά και υπάρχει πάντοτε η απειλή να ε, να διαφύγουν τα κεφάλαια από όπου υπάρχει υπερβολική ρύθμιση και γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ζακ Ντελόρ προχθές ότι ίσως πρέπει να δεχτούμε Πρέπει μάλλον να αντισταθούμε σε αυτή την ε, επιχειρηματολογία ότι είμαστε όμοιροι των χρηματαγορών όσο προς το που τοποθετούμε τα κεφαλαία μας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να σας πω πόσο όσοι είναι θύματα αυτών των κρίσεων χωρίς να ε, ε, φταίνε πρέπει να τονιστούν. Και θέλω να κάνω δύο δύο ερωτήσεις. Ξέρω ότι δεν ήταν μέσα σε αυτά που αναλάβατε να πείτε, αλλά ίσως επειδή ξεκαθαρίσατε πολλά πράγματα, μπορείτε να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε, διότι δύο φορές στο Κοινοβούλιο ψηφίσαμε ότι θα έπρεπε να, χρημα... Ε, να επιβάλλουμε φορολόγηση στις ε, χρηματικές συναλλαγές. Ε, η πρόταση αυτή μπορεί ίσως να απαντήσει εις ε, την πρόκληση την οποία εντοπίσατε και δεν υπολογίζουμε παρκώς διότι οι χρηματαγορές είναι πολύ περίπλοκες και με το παραμικρό οι υπεύθυνοι αλλάζουν, μια νέα, αλλάζουν τη στρατηγική τους αν επινοήσουμε κάτι νέο αλλά υπάρχει μια ιδέα η οποία δεν προέρχεται από τις χρηματαγορές και αποδεικνύει ότι μετά από αυτή την κρίση για πρώτη φορά θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε μία πρόταση και μία λύση η οποία δεν ανήκει στα μέσα και στα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι των κρίσεων. Πώς λοιπόν εσείς αξιολογείτε αυτή την πρόταση και πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να συνδυαστούμε με κινήσεις των υπευθύνων στην Αμερική για να προωθήσουμε μία τέτοια πρόταση. Δεύτερον, σχετικά με το G20 το οποίο νοσονούπο θα ξανασυνέλθει υπό Γαλλική Προεδρία. Και επανέρχομαι στο πρώτο μου επιχείρημα, ότι οι υπεύθυνοι των χρηματαγορών ε, δεν ε, μπορούν να λύσουν τα παγκόσμια προβλήματα, τα οποία όμως μπορούν να λυθούν σε επίπεδο G20. Τι μπορούν λοιπόν να κάνουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι για να χρησιμοποιήσουν αυτό το χώρο για να μην μοιάζει το μέλλον με το παρελθόν το οποίο διανύσαμε. Επιτρέψτε μου καταρχήν να κάνω μία παρατήρηση. Απαντώντας σε ερωτήσεις αυτές ε, μπορώ να σας πω ότι μπορώ να μιλήσω άνετα εν ονόματι της Επιτροπής μου και να παρουσιάσω τη δικιά μου άποψη. Αλλά όσο αναφέρεται σε αυτήν την ρυθμιστική διαιτησία, regulatory arbitrage ε, και θα προσπαθήσουμε να ε, μην να μην υπάρξει μια κίνηση μόχλευσης των μεν χωρών υπέρ ή κατά των άλλων για το πώς τα χρήματα μπορούν να κινηθούν, τα κεφάλαια να κινηθούν όπου επιλέξουν και να τοποθετηθούν εκεί και θα πρέπει η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, να εξασφαλίσουν ότι θα έχουμε ένα συνεπές ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μην είναι οι χώρες μας ε, όμοιροι των ε, προβλημάτων των πιο αδυνάμων διότι σας είπα ότι είμαστε, υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις αρχές της του 2000 όπου οι αμερικανικές το αμερικανικό κράτος είχαν, είχε καθορίσει δύο ρυθμιστές παρόλο που αυτή η οργάνωση δεν είχε κάποια προϋπηρεσία σαν χριστός διαχειριστής. Η δε AIG είχε μία επιτήρηση ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μία πιο στενή διασύνδεση μεταξύ των δύο στελεχών κατά τρόπον ώστε να υπάρχει καλύτερη εποπτεία. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι στην νομοθεσία Dodd Frank έγινε μία έντονη συζήτηση. Ε, δεν θυμάμαι ε, εάν υπερψηφίστηκε μόνο από τους δημοκράτες ή ψήφισαν και κάποιοι ρεπουμπλικάνοι αλλά είπαμε ότι εάν υπήρχε μία κατάρρευση ενός, μιας οργανώσεως θα έπρεπε η Federal Deposit Insurance Corporation δηλαδή η ομοσπονδιακή ασφάλεια να αναλάβει το κόστος Τη της διασώσεως και οι διατάξεις αυτές ισχύουν ακόμη και τώρα. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ο Πολ Ράιαν, ο πρόεδρος των, της ομάδος των Ρεπουμπλικάνων που ζητεί να καταργηθεί αυτό το σύστημα ενώ θέλαμε να υπάρχει μία εξασφάλιση για τα, τους υπερβολικούς κινδύνους που μπορεί να αναλαμβάνονταν. Θέλω όμως να σχολιάσω εδώ το θέμα. Ένα πολύ σοβαρό μέτρο που μας ανησυχεί είναι ότι το βασικό ρόλο συνεχίζει και τον παίζει η Wall Street, το Αμερικανικό χρηματιστήριο. Και βλέπουμε ότι και η δικιά μας ε, κυβέρνηση αλλά και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και οι ε, ε, εθνικές ευρωπαϊκές ε, κεντρικές τράπεζες συνεργάστηκαν. Δηλαδή όταν οι δύο εταιρείες Freddie May, Mac και Fannie Mae κατέρευσαν κανείς δεν το είχε προβλέψει και δεν είπε ότι δεν θα βοηθηθούν. Ευχαριστώ Φιλ και Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάινεν και στην κυρία ε, Κράτσα που εκπροσωπούν την ε, ομάδα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ε, για την πολύ καλή σας ανάλυση και την ε, εργασία σας την οποία ε, μας είχατε ήδη ε, παρουσιάσει σχηματικά όταν σας επισκεφθήκαμε στην Αμερική. Νομίζω ότι οι γενικές γραμμές των συμπερασμάτων σας συνάδουν με τα δικά μας συμπεράσματα στην Ευρώπη. Οπότε ίσως η πρώτη σας ανάλυση είναι σωστή. Δηλαδή ότι μπορεί να έχει αποφ Μπορεί να είχε αποφύγει κανείς αυτή την ε, ε, κρίση αλλά ε, η ύψιστη ευθύνη οφείλεται εις τους πολιτικούς και ουσιαστικά επί του θέματος αυτού υπήρξε κάποια πλήρης ρυθμιστική αποτυχία. Ε, τώρα λοιπόν και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ε, εργαζόμαστε με διαφορετικές μεθόδους και με διαφορετικούς τρόπους αλλά προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια ρυθμιστική διαιτησία και να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω έχετε επίσημες ή άτυπες προτάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ε, το G20 δεν ε, είναι πολύ δραστήριο για να αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η κυρία Κράτσα έχει τώρα το λόγο. I will speak Greek, ε, Mr. Χαίρομαι και εγώ πολύ που έχουμε την ευκαιρία, το προνόμιο σήμερα να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση της αποτίμησης των πορισμάτων της ε, Επιτροπής της οποίας προεδρεύατε για την αποτίμηση της κρίσης. Ε, χαίρομαι και ιδιαίτερα επειδή έχετε ελληνική καταγωγή και μάλιστα και από την ίδια περιοχή που είμαι και εγώ από τα Επτάνησα ε, κύριε Αγγελίδη, άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που μας παρουσιάσατε και πέρα από την αποτίμηση και τα πορίσματα και τις προσωπικές σας ε, προτάσεις ε, για τα βήματα που πρέπει να κάνουμε και μάλιστα σημείωσα με ιδιαίτερη προσοχή την πρόταση για τη συνεργασία μεταξύ ηνωμένων πολιτειών και ευρώπης οπωσδήποτε στο διεθνές παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η συνεργασία δύο μεγάλων οικονομικών δυνάμεων και χρηματοπιστωτικών αγορών όπως είναι η Ευρώπη και η Αμερική είναι αναπόφευκτο αναγκαίο και μάλιστα ακόμη περισσότερο σε επίπεδο G20 ε, προσπαθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσει την ανάγκη κοινών πολιτικών. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εάν ε, έχετε ασχοληθεί εσείς προσωπικά ή η Επιτροπή σας με, τις, ε, με τα κοινά σημεία ή τις διαφορές ε, των αντιδράσεων των δύο αγορών μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής ως προς τις συνέπειες της κρίσης και των αντιδράσεών τους για να κάνουν το, βήμα, το επόμενο βήμα της εξυγίανσης της ρύθμισης. Ξέρετε αυτό το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ δραστήριο από την πρώτη στιγμή να ζητήσει ρυθμιστικά πλαίσια εποπτείας και μάλιστα ήταν πιο τολμηρό και απαιτητικό από ό,τι και οι εθνικές κυβερνήσεις και τελικά ε, καταφέρνουμε να προχωρούμε όσο το δυνατόν και περισσότερο στην εποπτεία και την ρύθμιση. Ε, αυτό λοιπόν ήθελα να σα ρωτήσω η πρώτη με ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να πληρώσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι έχει συνηθίσει να πληρώνει ο τομέα, κυρίω τώρα που υφίσταται η κοινωνία και η οικονομία τι συνέπειε τη κρίση που προκάλεσε. Ε, διήστανται οι απόψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το φόρο, τι θα ήταν πιο κατάλληλο, ένα φόρο στι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ στην Ευρώπη μόνο εάν δεν επιτευχθεί διεθνή συμφωνία, μια φορολόγηση τύπου α, α, φόρου προστιθεμένης αξίας. Ήθελα να ρωτήσω αν και εσείς κάνετε τέτοιες σκέψεις και μελετάτε πιθανές περιπτώσεις στην Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όπου μου θυμίσατε ότι έχουμε κοινή κληρονομιά όπως όλοι όσοι έρχονται από τα θαυμάσια Επτάνησα Θέλω όμως ε, να σχολιάσω γιατί διάβασα όσο μπορούσα πώς αντέδρασε η Ευρώπη, τις πρωτοβουλίες που αναλάβατε και ουσιαστικά μπορώ να σας πω ότι και εμείς τι έχουμε κάνει στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, τον 1,5 τελευταίο χρόνο και βάσει των ε, ερευνών μου θα κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Ο καλύτερος τρόπος των νομοθετών κατά τη γνώμη μου είναι να υπάρχουν πολύ περισσότερες διμερείς συζητήσεις μεταξύ των ρυθμιστών διότι υπάρχουν ε, συστημικά θέματα που τίθενται αλλά υπάρχουν και θεσμικά θέματα ε, θέματα των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων διότι αυτό που ήταν ε, πολύ καλό ήταν ότι είδα πως οι επενδυτικές τράπεζες συνεργαζόντουσαν με τους επιτηρητές τους και πόσο διαμορφώθηκε ε, ε, μετά το 2004 η συνεργασία που δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι και αν κοιτάξετε την AIG και την ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία θα δείτε το γραφείο του επιτηρητή θα πρέπει να επιβλέπει όλη την εταιρεία, όλη την AIG ας πούμε, όχι μόνο το ταμιευτήριο δεν είναι δυνατόν δηλαδή ο, ε, ένα, ε, μια οργάνωση να υπογράψει ε, ε, μία συμφωνία χωρίς να έχει ρωτήσει τη μητρική όπως μας είπε και χωρίς να γνωρίζει ε, ποιες ήταν οι ευθύνες που είχαν αναρριφθεί για τα credit default swap της AIG και για την κατάρρευση η οποία τελικά οδήγησε σε μία διάσωση ύψους 180 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Πρέπει λοιπόν η επιτήρηση αυτή να είναι διασυνοριακή και οι οργανώσεις επιτηρήσεως να είναι διασυνοριακές. Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές θέλω να πω το εξής. Έχω προσωπικές απόψεις και πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε κατά κάποιον τρόπο ε, ως εξής. Πρέπει στην Αμερική, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά το κοινό θεωρεί ότι είναι ένας προσεκτικός ασφαλιστής. Ε, και ε, είδαμε ότι όποιος κατέρευσε διεσώθη ο σωστός λοιπόν ασφαλιστής θα πρέπει να σας προστατεύσει να μην σας αφήσει να πηδήξετε από το αεροπλάνο χωρίς ε, ε, να φοράτε ένα λεξίπτωτο και να εξασφαλίσει ότι έχετε συγκεντρώσει επαρκή αποθέματα. Στην Αμερική είχαμε ένα αρκετά καλό σύστημα όσον αφορά την Federal ε, ε, ε, Deposit Insurance Corporation όπου επιβάλαμε μία πληρωμή εις τις διάφορες οργανώσεις ώστε να καταρτήσουμε θέματα. Θεωρώ λοιπόν προσωπικά ότι πρέπει να υπάρξει ε, κάποια επιβολή συνδρομής ώστε να καλύπτονται οι κίνδυνοι σε περίπτωση μιας κατάρρευσης. Δεν μπορώ να μιλήσω εδώ για τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει το σύστημά σας, αλλά μπορώ να σας πω ότι τώρα στην Αμερική έχουμε ένα ε, νέο προπολογισμό που κατέθεσε ο Πολ Ράιαν για το προϋπολογισμό πέραν του 2012 οπότε δεν θα είναι δυνατόν να ε, ε, καταβάλει κανείς αυτό το ποσό που θα έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται σαν απόθεμα και αυτό θα είναι καταστροφικό. Υπάρχει και άλλη μια συζήτηση στις Ηνωμένε Πολιτείες πώς το, το, οι τόκοι ε, για τα διάφορα ταμεία και τα ομόλογα πρόκειται να καταβάλλονται αν θα φορολογούνται ε, διότι εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κεφαλοχικά κέρδη είναι ε, φυσιολογικό κεφάλαιο το οποίο έχει κερδιθεί και άρα δεν ε, ε, χρειάζεται να μην ε, περιληφθεί ο κύριος Πρεσέρο. Ο κύριος Κομφεράτη πρώτος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθηγητά Αγγελίδη, χρησιμοποίησατε εσείς λόγια πολύ ξεκάθαρα και σταράτα για να παρουσιάσετε τα συμπεράσματα της Επιτροπής της οποίας προεδρεύσατε. Κάποιες κρίσεις σας παρουσιάσατε και κατά άποψή μου κάποιες κρίσεις σας είναι ιδιαίτερα εκτιμήσιμες, αξιέπαινες, διότι έχουν την εικόνα της ειλικρίνειας. Είπατε ότι η κρίση ήταν προβλέψιμη. Και εκείνο με έπληξε πολύ. Διότι έτσι υπονοείται και αναγνωρίζεται θα έλεγα στην Επιτροπή σας και η Επιτροπή σας αναγνώρισε ότι από πλευρά πολλών φορέων της χρηματοπιστωτικής πολιτικής της Αμερικανικής κατά κάποιες περιπτώσεις υποτίμηση και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έλλειψη, ξεκάθαρη έλλειψη ευθύνης που αυτά παρήγαγαν πρώτα τη φούσκα, την οικονομική, την κερδοσκοπική και μετά τις καταστροφικές συνέπειες που μας παρουσιάσατε. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα υποπτίας ήταν πολύ αδύναμο, ίσως ιωνίων ύπαρκτων. Φαντάζομαι ότι θέλετε να πείτε ότι και στο μέλλον για να αποφευθεί επανάληψη τέτοιου είδους φαινομένων είναι απαραίτητη όχι μόνο η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας αλλά πιθανότατα και ε, μια, να γίνουν πιο αυστηρές οι, οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε άτομα ή σε φορείς που υπολείπονται των ευθυνών τους, δεν ανταποκρίνουν τις ευθύνες τους. Αυτό με εκπλήσει πάρα πολύ, διότι στη χώρα σας όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια διαδίδεται η πρακτική της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και κυρίως οι τράπεζες ήταν οι πρώτες που χρησιμοποίησαν αυτού του είδους τη μέθοδο, αυτά τα εργαλεία. Όμως, μετά από αυτό που συνέβη, είναι προφανές ότι μεταξύ της περιγραφής της συνοχής και της ηθικής και από τη μία και των συγκεκριμένων πράξεων υπάρχει μια άβυσος μεταξύ των δύο. Διερωτώ με μήπως θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε το δεχόμενο συστήματος πρακτικής κοινωνικών ευθυνών που θα συνοδεύεται όχι μόνο από την υποχρέωση να θετηθούν τα μέτρα, αλλά και από πολύ ισχυρές αυστηρές ε, κυρώσεις. Δεύτερο ερώτημα που έχω είναι το εξής. Είπατε εσείς ότι ίσως οι ζημιές αυτής της κρίσης θα διαρκήσουν, θα διαρκήσουν τουλάχιστον για μια γενιά οι ζημιές. Πιστεύω κι εγώ υπό το φως αυτών που επαληθεύσαμε και είδαμε και στη δική μας Επιτροπή ότι οι ζημιές είναι βαθιές και θα κρατήσουν πολύ καιρό και σε αυτό το μέρος του κόσμου. Λοιπόν, γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείες αποφάσισαν να εμπιστευθούν σε μια, σε μια επιτροπή που ασχολείται μόνο με τη χρηματοπιστωτική πτυχή της κρίσεως. Αν οι ζημιές για εκατομμύρια άτομα διαρκέσουν τόσο χρόνο, γιατί να μην ενταχθεί αυτή η επιτροπή μαζί με μια, σε μια άλλη επιτροπή ή να δοθεί άλλη εντολή σε αυτή την επιτροπή ώστε να εξετάσει και οικονομικές πτυχές μαζί και τις κοινωνικές πτυχές. Μας εξέπληξε το ότι είδαμε εμείς την Αμερικανική κυβέρνηση να θεσπίζει νόμους για την υγεία, δηλαδή να εισάγει ένα μηχανισμό πρωτοφανή του welfare state με όλες τις δυσκολίες που δημιούργησε και επιτάχυνε τα προβλήματα και δεν έλαβε υπόψη την παρέμβαση υπέρ των ατόμων εκείνων που είχαν πληγεί από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω να σε ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και για τα συμπεράσματα που μας παρουσιάσατε και που αναφέρονται παρόμοια συμπεράσματα και στον τύπο στην Ευρώπη. Το πρώτο συμπέρασμα που συναγάγατε ήταν ότι ήταν η κρίση που κάτι που μπορούσε να αποφευθεί. Δεν ήταν μοιραίο γεγονός, ήταν αποτέλεσμα αποτυχίας του συστήματος και για τους ιδιωτικούς φορείς αλλά και από πλευράς των δημοσίων φορέων. Κυρίως σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχε έλλειψη νομιμότητας όσον αφορά την ε, δραστηριοποίηση του δημόσιου τομέα και σωρεύτηκαν τα προβλήματα τα πράγματα πήγαιναν καλά. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο ε, να, άμα ακούγεται κόδων κινδύνου να τον πάρουν κανείς τα σοβαρά όταν βγαίνει χρήμα, τα πράγματα πηγαίνουν καλά και επικρατεί εφορία, είναι δύσκολο να σκέφτεται κανεί την καταστροφή. Άρα θα ήταν καλό να προλαμβάνονται αυτά τα προβλήματα. Ε, και σημειώσαμε ότι είπατε ότι υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα, διότι δεν υπήρχε ένα σαφέ όραμα σχετικά με αυτά που συνέβαιναν στο χρηματοδοτικό σύστημα. Και υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία θα ήθελα να σα θέσω και θα ήθελα να ακούσω ποιε είναι, ποιες είναι οι σκέψει σα πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα το χρέο. Ε, σίγουρα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό θέμα διότι το χρέος δεν είναι μόνο που αφορά τους ιδιώτες και τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την αξία των αγαθών, των στοιχείων ενεργητικού, των αξιογράφων για τη λειτουργία της ε, οικονομίας. Πρέπει να τεθούν όμως ε, κάποια όρια στις πιστώσεις. Λοιπόν, θα ήταν πιο χρήσιμο να περιγραφεί ε, σαφές... Το δεύτερο θέμα είναι αυτό το σύστημα των αμοιβών, των πριμ, γιατί υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι κάνουμε άλλα αντάλλον Πέρασε, λένε η κρίση, αλλά ακόμα γίνονται τα ίδια λάθη, λένε. Θα πρέπει πιο αποτελεσματικά να γίνεται η διαχείριση. τι γίνεται με την πιστοληπτική αξιολόγηση και τις σχετικές εταιρείε. Θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι είδους δείκτες, κάποιοι είδους σήματα, μηνύματα στους επενδυτές. Δεν πήγε καλά το σύστημα. Ούτε διάγνωση γινόταν, είχαμε συγκρούσει συμφερόντων. Θα πρέπει αμερόληπτα να λειτουργεί το σύστημα. Θα πρέπει σε βάθος να κάτσουμε και να δούμε το μοντέλο το οποίο ισχύει, αν πάσχει ή όχι. That's a lot. πολλά, πολλά με ρωτήσατε να δούμε αν μπορώ να μαζέψω τα διάφορα κομμάτια. Λοιπόν, το θέμα του κατά πόσο ήταν κάτι που μπορούσε να αποφευθεί η κρίση. Σε κάποιο επίπεδο φαίνεται απλό, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό, σημαντικό, είναι και μου σημασία, διότι αυτοί που θέλουν να ξεπεράσουν την κρίση, που τη χαρακτηρίσανε σαν μια ανομαλία μικρή στο δρόμο, παίρνουν μια θέση και λένε ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την κρίση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτή είναι η βάση για να μην δοθεί κάποια απάντηση και να μην θεσπίζεται κάποια πολιτική. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι εξεπλάγει. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία με καλή γνώση του χρηματοστικού τομέα. Αυτό θεωρούσα. Και εξεπλάγει από το επίπεδο των κοδώνων συναγερμού που χτυπούσαν, από τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες, για εκείνους που διαμορφώναν την πολιτική και για τους διάφορο, διάφορα ανώτερα στελέχη ε, των επιχειρήσεων που είχαν καθήκοντα και χρέη εναντί των μετόχων. Η έλλειψη δράσης λοιπόν έναντι πολύ σημαντικών πληροφοριών, ουσιαστικών πληροφοριών ήταν κάτι που με συγκλώνησε. Δεν νομίζω λόγω των σκοτεινών αγορών ότι καταλάβαινε ο κόσμος πολύ καλά ότι όταν έσκασε η στεγαστική φούσκα το πόσο μεγάλο και βαθύς ήταν ο αντίκτυπο. Αλλά σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλέ πληροφορίε για τις πρακτικές δάνειοδότησης, πολλέ πληροφορίε για το μέγεθος τη φούσκας της στεγαστική, για την πλήρωση των διαφόρων, ε, για τι γινόταν με τις ασφαλεί κλπ. Διερωτώ με, λοιπόν, εν ώψη όλων αυτών, γιατί δεν έγινε τίποτα. Διότι έτσι θα καταλάβουμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα το σύστημα αποζημιώσεων ήταν τόσο κερδοφόρο για να γίνεται η συναλλαγή χωρίς να βλέπει κανείς τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που ακόμα και εν ώψη πληροφοριών για επικείμενη, επικείμενο τέλος αυτού τέλος, επικείμενο τέλος της φυσαλίδας, εξακολουθούσαν να γίνονται συμφωνίες διότι έπαιρναν μεγάλη αποζημίωση τώρα ε, χωρίς να βλέπουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Στη Wall Street ε, έλεγαν IBG, YBG, δηλαδή αν φύγουν ε, όλα θα φύγεις και εσύ. Δηλαδή το σύστημα αποζημίωσης ήταν ο μεγάλος ηγέτης. Ε, αγνοήθηκαν τα σήματα προειδοποίησης, τουλάχιστον στη χώρα μας. Γιατί θεώρησαν ότι μπορούν να αυτοδιορθώνονται οι αγορές, ότι η αποτελεσματική αγορά λειτουργούσε και ξεπερνούσε τα πολιτικά κόμματα, διαμόρφωνε τις αποφάσεις της κυβερνήσεως και της κυβερνήσεως Μπούς και υπήρχε υπεποίθηση και μάλιστα μέχρι τέλος του 2007 άντε και κατά διάρκεια του 2008 υπήρχε το συνέστημα ότι οι αγορές θα διορθώναν τα προβλήματα από μόνες τους. Αυτό που δεν υπολόγισαν ήταν ήταν ε, το θέμα των αποσμιώσεων, οι πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες για να λαμβάνονται και πιο βασικές αποφάσεις και υπενοείται ότι η αγορά θα ακολουθούσε οθολογική προσέγγιση. Μας είπε ένας καθηγητής το εξή. Ο, ο νόμος της βαρύτητας πάντα ισχύει. Ε, ε, Η ιδεολογία δηλαδή λειτουργούσε σαν νόμο ότι η ελεύθερη αγορά μπορεί να λειτουργεί και να διορθώνεται η κατάσταση από μόνη τη. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα αλλάξει γρήγορα. Και ήταν ένα θέμα δυνατοτήτων. Δηλαδή, ταλέντο, ικανότητε από τη μια πλευρά, ότι έτσι μπορούμε να το κάνουμε, και ευελιξία, ταχύτητα με την οποία κινείται η Wall Street από τη μια και τη δυνατότητα που είχαν οι φορεί εποπτεία. Και η δυνατότητα τι, από τι διακρίνεται, από πολιτική βούληση, τότε βασίλευε η νοοτροπία πολιτική ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώ αυστηρό την εφαρμογή των νόμων. Αν διαβάσετε αυτό το, βιβλίο, περιέχει διάφορα που έλεγαν οι θυμιστικοί φορεί. Βλέπετε ότι οι υποπτικοί φορεί δεν έβλεπαν τη δουλειά του σαν προσπάθεια επιβολή και συγκράτηση των τραπεζών, αλλά να, λειτουργούν σαν ε, σύμβουλοι ε, των ε, τραπεζών. Μίλησα με τον πρόεδρο Μπεν Μπερνάκη για το θέμα αυτό. Δεν υπήρχε ούτε βούληση ούτε δυνατότητα να το κάνω αυτό. Δηλαδή, ήταν θέμα πώ να προσεγγίσει κανεί ταλαντούχου γνώστε στο δημόσιο τομέα, να του κρατήσει, διότι υπήρχε έλλειψη αντιστάθμιση μεταξύ αυτά που ήθελε η Wall Street από τη μία με αυτά που ήθελαν οι θρησκευτικέ αρχέ από την άλλη. Άρα συμπληρώθηκε από ένα άλλο φαινόμενο η όλη κατάσταση. Ο ιδεολογικό παράγων ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα επιστρέψω στον Άλαν Greenspan. Υπήρχαν και άλλοι, αλλά να επιστρέψω στον Greenspan. Όταν επανειλημμένα του έδιναν πληροφορίε για του κίνδυνου που έπαιρναν οι δανειοδότε όσον αφορά τα δάνεια και κάθε φορά έτεινε να μην επιβάλλει συμπληρωματικού όρου και είπε μάλιστα σε εμά ιδιωτική συνομιλία που είναι δημόσια τώρα και θέσιμη στο διαδίκτυο είπε ότι όπου βλέπετε πάρα πολύ έτσι, εύκολες δανειοδοτικές πρακτικές, δεν χρειαζόμαστε περισσότερες ρυθμίσεις εκεί, αλλά επιβολή του ήδη υπαρχόντος νόμου. Όταν είδαμε λοιπόν εμείς από τα αρχεία ότι μεταξύ του 2000 και του 2006 η περίοδος κατά την οποία είχατε τις πιο εξωφρενικές πρακτικές δανειοδότησης που εφαρμοζόταν στη χώρα μας και βλέπατε ότι η Federal Reserve παρέμπεψε μόνο τρεις υποθέσεις άδικη αθέμητης δανειοδότηση στο Υπουργείου Δικαιοσύνη προ έρευνα. Δύο μικρές τράπεζες, μία στο Ελληνόη και μία στην Καλιφόρνια και, ε, και το υποκατάστημα της Νέας Υόρκης της Practice ε, General. Πίστευαν, λοιπόν, έλλειψη διόρθωσης των κινήσεων των αγορών, έλλειψη δυναμικότητας, η, δυνατό, η δύναμη του χρηματοδοτικού τομέα μας εμπόδισαν να λάβουμε δράση και όλα αυτά είναι πολύτιμα μαθήματα. Το θέμα αυτό της αποτροπής είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε. Δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Ε, πολλοί με, τα, με τη συμπεριφορά τους έφτασαν στα όρια. Τα όρια δηλαδή της διοντολογικής σωστής συμπεριφοράς που δεν μπορεί να εφαρμόζεται αν θες να έχεις μακροπρόθεσμα βιώσιμη οικονομία. Και υπήρχαν και εκείνοι που πέρασαν τα όρια και υπέστησαν ελάχιστες κυρώσεις, όπως η Citigroup, παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια όλου του 2007, η Citigroup Όσον αφορά το επενδυτικό κοινό, έλεγε ότι η έκθεσή της στα subprime mortgages ήταν περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουμε νόμους στη ΣΥΠΑ, δεν ξέρω ε, ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί νόμοι. Οι δικοί μας νόμοι απαιτούν έγκαιρη και ακριβή αποκάλυψη προς τους μετόχους και προς το επενδυτικό κοινό των πληροφοριών. Κάπου το καλοκαίρι του 2007, η ηγεσία της Citigroup καταλαβαίνει ότι η έκθεση είναι ακόμα μεγαλύτερη διότι είχαν και διάφορες φορείς που ήταν εκτός του ισολογισμού τους. Το Σεπτέμβριο η έκθεση είναι από 50 δις δολάρια και πάνω και 15 Οκτωβρίου η Group, το Διοικητικό Συμβούλιο της City Group και η Επιτροπή Ελέγχου του Κινδύνου παίρνουν λεπτομερέστατη έκθεση, την πήραμε και εμείς, όπου εκεί αναφερόταν ότι παρά αυτά που δημοσία παρουσιαζόταν, η Citigroup είχε περίπου 55 δισεκατομμύρια δολάρια έκθεση σε subprime στεγαστικά δάνεια. Την ίδια μέρα λέει στο επενδυτικό κοινό η Citigroup για μία ακόμη φορά ότι είναι στα 13 δις. Πέρασαν και τέσσερι εβδομάδε για να πούν την αλήθεια. Ποια κύρωση του επευλήθη. Ο αρμόδιο υπεύθυνο έβγαλε 7 εκατομμύρια δολάρια το 2007 και πλήρωσε πρόστιμο 100.000 δολάρια. Ένας άλλος που έβγαλε 3 εκατομμύρια ε, έφαγε ένα πρόστιμο με 5.000 ε, δολάρια. Πού είναι το αποτρεπτικό της ποινή, το να έχει αριθμιστικό καθεστώ με πραγματικά αποτρεπτικά μέτρα είναι πολύ σημαντικό. Ήταν η βάση ε, του ρυθμιστικού καθεστώτο μετά τη μεγάλη ύφεση στο... στη ΣΥΠΑ. σω να πω κάνα δύο άλλα πράγματα. Δεν πρέπει να, περιγράψω του διάφορου φορεί ε, βαθμολόγηση πιστοληπτική ικανότητα, που είναι ανίκανοι και δείχνουν κατακαιρματισμένη εικόνα. Είναι σπασμένο το ε, μοντέλο. Πληρώθηκαν από εκείνου που ήθελαν να πάρουν ε, την διαβάθμιση τριπλό Α δεν είναι βιώσιμο το μοντέλο. Υπήρχαν κάποιε ρυθμιστικές αρχέ στι ΗΠΑ, αλλά δεν έφτασαν στο βαθμό που θα θέλαμε. Για πρώτη φορά οι υπηρεσίε βαθμολόγηση πιστοληπτική ικανότητα ε, δεσμεύονται περισσότερο από την αρμόδια επιτροπή τώρα. Πρέπει να αποκαλύπτουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούν, τι ανάλυση κάνουν. Και αυτό που θα σα εκπλήξει, αν το δείτε αυτό, θα είναι που ανέφερα την Moody's. Να μην πω την Standard Poor's που ήταν ε, κάναμε έρευνες συγκεκριμένων υποθέσεων. Η Moody's λοιπόν, σας είπα, 45.000 ε, τίτλους από το 2007 θεώρησαν τους φορείς αυτούς σαν τριπλό α. Δεν είχαν κανένα μοντέλο για να αναλύσουν ε, τα, τη δανειοδότηση των subprimes του 2006. Είχαν βασιστεί σε ένα παλιό μοντέλο του 1996 που αναπτύχθηκε από prime mortgages Οπότε πρέπει να αποκαλύψουν τώρα ποια είναι τα μοντέλα που χρησιμοποιούν. Στο τέλος όμως εγώ πιστεύω προσωπικά ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από ένα σύστημα όπου εκείνοι που εκδίδουν ε, τα αξιόγραφα πληρώνουν για την βαθμολόγηση και να, οι επενδυτέ να πληρώνουν. Οπότε υπάρχει αλλαγή συμφερόντων. Ο γερουσιαστή Αλ Φράγκλιν έκανε μια πρόταση που συμπεριλήφθη στον νομοσχέδιο Dodd Franklin όπου εκεί θα απαιτείται μια μελέτη για να δούμε αν μπορούμε να μετακυθούμε σε ένα σύστημα όπου να υπάρχει μια επιτροπή που θα διαλέγει το φορέα βαθμολόγηση και όχι η Goldman να διαλέγει ποια θα είναι η υπηρεσία που θα κάνει βαθμολόγηση ή κάποιο άλλο να διαλέγει το δικό του φορέα βαθμολόγηση πιστοληπτική ικανότητα. Το θεμελιώδε μοντέλο ήταν διεφθαρμένο, ήταν στραβό. Δεν ξέρω πώ αλλιώ να το πω. Α, και άλλο ένα ερώτημα και το επίπεδο του χρέους. πιστεύω, κατόπιν σκέψεως, ότι θα ήταν συνε... θα έπρεπε να είμαστε συνετοί όσον αφορά τα πρότυπα και τα χρέη. Προέρχομαι από αυτόν τον τομέα, εξεπλάγην το 2006, όταν ξαναμπήκα στο ιδιωτικό τομέα, αφού έφυγα σαν αρμόδιος οικονομικά της πολιτείας της Καλιφόρνια. Περισσότερο από τη μισή μου ζωή την πέρα στο ιδιωτικό τομέα. Επέστρεψα το 2007, αρχές του 2007 και εξεπλάγην, βλέποντας ότι οι μπορικοί φορείς έπαιρναν 95% και 100% χρηματοδότηση για ε, αξίες που ήταν υπερτιμημένες και οι θεσμοί που έδιναν ε, τα δάνεια ε, ήταν πολύ στηριγμένοι. Οπότε πρέπει να υπάρχουν πρότυπα που εφαρμόζονται και να είναι λογικά τα πρότυπα. Να εκφράσω με τελική σκέψη. σω θα τα σταματήσω εδώ μακριγόρισα κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, θα πρέπει να προσέχουμε και το χρόνο. Έχουμε ένα μισάωρο μπροστά μα και έχω κατάλογο έξι συναδέλφων. Τώρα που το είπατε, 30 δευτερόλεπτα λοιπόν. Υπάρχει ένα καλό μοντέλο που ίσως θα έπρεπε να εξετάσετε. Το Community Reinvestment Act για την κοινωτική επαναχρηματοδότηση του ΣΥΠΗΝ. Μπορείτε να το σκεφτείτε. Οι τράπεζες δανειοδοτούν και δίνουν δάνεια σε γειτονιές που δεν δανειοδοτούσαν, σε φτωχ... δανειοδοτούν φτωχές γειτονιές τώρα, που έπρεπε να ταιριάζει και με προϋποθέσεις για ασφάλεια. είναι ένα μοντέλο ε, κοινωνικής ευθύνης που στεριάζει μαζί με την ανάληψη του σωστού κινδύνου. Πρόεδρος, κανονικά η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα, οι φιλέθεροι και οι δημοκράτες θα έπρεπε να παρέμβουν, αλλά θα δώσω το λόγο στον Γκέι Μίτσελ, διότι ξέρω ότι ίσως δεν μπορεί να μείνει μέχρι το τέλος της σα και μετά θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Ο Γκέι λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιλίδη. Πόσο ελεύθερε είναι οι αγορέ, στοιχειώδη ερώτηση. Τώρα, πάνω σε αυτό επίσης μιλάμε για ελεύθερα ΜΜΕ και ξέρουμε ότι ολόκληρη το μίσος, τα κομμάτια αυτού του κλάδου είναι εξαρτημένα. Εμείς τα λέμε, οι βουλευτές, ότι πολλές φορές αυτά τα ΜΜΕ ε, διαπλέκονται. Πολλά, πολλά, ολόκληρα κομμάτια των μέσων ενημέρωσης του κλάδου των μέσων ενημέρωση και θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ε, αυτό υποτίθεται. Οπότε θα έπρεπε να μην υπάρχουν τέτοιου διαπλεκόμενε συμφέροντα. Γι' αυτό σα λέω ότι κατά τη γνώμη μου η δημοκρατία εδώ έχει αποτύχει. Και σε πολιτικό επίπεδο και σε επιχειρηματικό. Οι εταιρείε σέβονται τους μετόχους τους. Για πες μας επομένως, υπάρχει ελευθερία στις αγορές. Μπα και χειραγωγούνται από αυτού που εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι υπέρ τη ελεύθερη αγορά, αλλά θέλω να είναι αυθεντικά, πραγματικά ελεύθερη αγορά και να μην ελέγχεται από κάποιου οι οποίοι τι χειραγωγούν. Οφελούνται, κερδίζουν οι λίγοι. Χειραγωγούν την αγορά. Το έχετε μελετήσει το θέμα. Πόσο ελεύθερη είναι η αγορά. I think it's fair to say we probably, <sighs> you know, we had a year and a half. That's a very big question. I will say this. We did. Ναι, ναι, κρεμούσε το θέμα εδώ. Το μελετήσαμε 1,5 χρόνο. Κάτσαμε και κοιτάξαμε τι στοιχεία έχει η Επιτροπή Χρηματιστηρίου. Αυτοί οι ισχυρισμοί, αν στέκουν. Αυτό το τεχνητό φούσκωμα των τιμών να δούμε δηλαδή, έχουν δει περιπτώσεις όπου κάποιοι χρηματιστές διαμορφώνουν τεχνητά τις τιμές και προέκυψε ότι όπως έχει σήμερα η δομή της αγοράς διοικητικά συμβούλια, ε, μετοχές. Ε, δεν, λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Και εγώ ήμουν σε διοικητικό συμβούλιο. Σε, στο μεγαλύτερο συνταξιδοτικό ταμείο. Στο πρώτο και στο δεύτερο συνταξιδοτικό, τα μεγαλύτερα ταμεία. Ήμουν στο διοικητικό συμβούλιο εκεί. Ταμείας. και πασχίζαμε για να δούμε τι γίνεται με τη συμμετοχή μας στο, στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρεών. Και βλέπαμε ότι η δημοκρατία στην οποία διαμορφώνεται η πολιτική της εταιρείας από την πλειοψηφία των μετόχων είναι ένας μύθος σε πολλές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μετόχων και δεν γινόταν. Δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Γι' αυτό σας λέω. Διαβάστε την έκθεσή μας και θα δείτε. Δυσλειτουργούσαν οι εταιρείε. Και πολλά τα οποία έκαναν αυτές τις εταιρείε δεν τα ξέρανε οι διευθυντές σύμβουλοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τα κορυφαία λέει ότι μιλάγαμε για 79 δις ανοίγματα για την Goldman Sachs. στη διακυβέρνηση. Ήταν, ήταν κάποιες ομάδες μικροί θύλακες, ας το πούμε, κάποιων στελεχών που κράταγαν τα ενία. Στο Warren Buffett. Ο Warren Buffett τι έκανε, πήρε το 20% του Μούντις και με άλλους τρεις είχε την πλειοψηφία πάνω το 50%. Όλα αυτά χωρίς να ξέρει καν πού είναι τα γραφεία. Ε, δεν είναι αυτό πρότυπο, δεν είναι αυτό υπόδειγμα, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση για τη διακυβέρνηση. Δεν είναι ένα πρότυπο παραγωγής επένδυσης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Όλε Μήτρο, συνάδελφό μας από την Σουηδία, δεν μπορεί να παραστεί. Είχε κάποια υποχρέωση ε, στο κόμμα του. Οπότε, ανταυτού, θέλω να σας πω τα εξή. Τρία την. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε τρία θέματα. Πρώτον, μιλήσατε για το αλόμπις στην Ουάσιγκτον και κάθε φορά που διαβάζω τους αριθμούς ε, εντυπωσιάζομαι ότι χρειάζεται κανείς να συγκεντρώσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να γίνει υποψήφιος για πρόεδρος και χρειάζονται εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια για να ε, ε, μπορέσει κανείς να γίνει γερουσιαστής ή βουλευτής. Άρα ε, μιλάμε για πλουτοκρατία, όχι για αριστοκρατία. Λοιπόν, ε, ο οικονομικός τομέας επίσης τώρα αντιπροσωπεύει το βάρος της οικονομίας ε, που είναι πάρα πολύ υψηλών. Και το ερώτημα μου είναι, υπάρχει κάποια κίνηση ή κάποια πρόθεση να αποβιομηχανοποιηθεί η ε, αμερικανική βιομηχανία για να επαναφέρουν στην Αμερική ορισμένες βιομηχανίες. Επίσης, ε, έχουμε ένα πρόβλημα στην ε, Ευρώπη και εσείς έχετε το δημόσιο χρέος στην Αμερική. Πόσο ποσοστό του δημοσίου χρέους οφείλεται στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις. Ε, σήμερα όντως με προκαλείτε πνευματικά. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να σας απαντήσω εξαιρετικά. Ε, διότι στην έκθεση μας νομίζω ότι αναφέραμε ότι η βιομηχανία των οικονομικών ε, υπηρεσιών δαπάνησε 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο κυβερνητικό. Ε, δεν έχουμε περιλάβει ε, τα ποσά από το 1999 έως το 2008 ήταν 2 δισεκατομμύρια δολάρια το, το ποσό που δαπανήθηκε χωρίς τους συμβούλους. Και εγώ προσωπικά, ε, επειδή έχω υπάρξει εκλεγμένος εκπρόσωπος στη χώρα μου, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ανισομερής η κατανομή. Υπάρχει ε, μεγάλη επιρροή, μεγάλη ισχύς και ο οικονομικός τομέας είναι στο επίκεντρο του διαλόγου για τα οικονομικά. Είναι πιο σημαντικό και από τις συνδρομές για την προεδρική προεκλογική εκστρατεία. Ε, βλέπουμε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών, οι Treasure Secretaries προέρχονται από τον εξοκοινοβουλευτικό χώρο και ε, η κατάσταση αυτή οφείλεται σε ορισμένους λόγους. Ένας λόγος αναφέρεται στο ανώτατο δικαστήριο διότι το 1976 μετά το Watergate και την πτώση του Νίξον υπήρξε ε, μία νομοθεσία η οποία υπερίσχυσε και περιόριζε το ποσό ανά άτομο για συνδρομή σε προεκλογική εκστρατεία ε, και ε, ε, το, το, τίμημα ήταν ο εις της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης. Δηλαδή ο, η νομοθεσία αυτή δεν μπόρεσε να περιορίσει τις δραστηριότητες των τρίτων που δεν είχαν άμεση σχέση με τον υποψήφιο και ε, τώρα ε, περιορίζονται με τα κόμματα για τα χρήματα που μπορούν να συγκεντρώσουν ενώ τα άτομα ε, δεν περιορίζονται για την προσωπική τους προεκλογική εκστρατεία και τελευταίως το δικαστήριο πρόσθεσε ορισμένα μέτρα υπάρχουν αποφάσεις που επιτρέπουν σε εταιρείε που δύσκολα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ομοσπονδιακό επίπεδο να προτείνουν ή να αντιδράσουν σε έναν υποψήφιο οπότε ορισμένα ποσά θα μειωθούν στο μέλλον. Όταν ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ μου έκανε εντύπωση η εργασία της Επιτροπής Κρίσεως εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο διότι εσείς ε, εστιάζεστε στην διάγνωση και στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να είναι ανταγωνιστική, τι επενδύσεις χρειάζονται και πιστεύω ότι στη χώρα μας αυτό είναι ένας χώρος όπου έχουμε έλλειμμα πολιτικής, όπου δεν προσέχουμε επαρκώς τα μέτρα που πρέπει να αναλάβουμε για να έχουμε προϊόντα υψηλή υψηλής ποιότητος και να πληρώνουμε παρκείς μισθούς. Αυτό είναι ένα έλλειμμα στη χώρα μας και ε, είμαι υπεύθυνο της Apollo Alliance ε, όπου υπάρχουν ε, εργοδοτικές οργανώσεις και επικεφαλής κοινωνικών κινημάτων για να καταρτήσουμε μια οργάνωση όπου μπορούμε να ηγηθούμε για τις ανανεώσιμες θα κάνουμε πηγές ενεργείας, όχι μόνο ηλιακή αλλά και άλλες και ε, προσπαθούμε ε, να ε, καθοδηγήσουμε την ζήτηση, θα προσπαθούμε να υπάρξει κίνηση σε, και παραγωγή σε εθνικό επίπεδο και βλέπω ότι και εσείς ασχολείστε με το τον ίδιο τρόπο με το χώρο σας. Ναι. Ε, το, μετά, η επιρροή της κρίσεως στο δημόσιο χρέος. Παρόλες τις ε, ε, αιτιάσεις της δεξιάς, πιστεύω ότι η κρίση επηρέασε πάρα πολύ τον ομοσπονδιακό ο προπολογισμό λόγω της μειώσεως των εισοδημάτων μπορώ να μιλήσω για την Καλιφόρνια και να σας δώσω ένα παράδειγμα διότι η κρίση επηρέασε πάρα πολύ τα δημόσια, τις δημόσιες δαπάνες και το χρέος διότι η Καλιφόρνια για στις καλές της μέρες ήταν πάντοτε ε, ε, εξόδευε περισσότερα από ό,τι συγκέντρωνε. Ε, όταν είχα ήμουν υποψήφιος ε, εναντίον του Σουάρτσενέγκερ το 1996 για κυβερνήτη. κυβερνήτης είχα εκφράσει την ανησυχία για την πολιτεία μας αν υπήρχε ε, κατάρρευση των οικονομικών. Αυτή ε, τη στιγμή έχουμε 260 δισεκατομμύρια έλλειμμα με έναν προπολογισμό πληθυσμό 80 δισεκατομμυρίων. Ε, υπάρχει μία πτώση σήμερα και οφείλεται αυτό εις ε, την ε, μείωση της παραγωγής, της κατανάλωσης και των, των ποσών τα οποία διαπιστώσαμε τελευταίως. Βλέπετε ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση, έχει μειωθεί η παραγωγή, όλα είναι πεσμένα. Και ε, ε, πρέπει να σας πω ότι ο μέσος ε, δάσκαλος στο Wisconsin έχει, ε, ε, έχει 50.000 ευρώ το χρόνο και η μέση σύνταξη στην Καλιφόρνια για εκπαιδευτικό είναι 2.400 δολάρια. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, θα συνεχίσω πάνω σε αυτά που ρώτησε ο κύριος Κλίντς για το παράδειγμα της Καλιφόρνιας. Λοιπόν κύριε Αγγελίδη, ποια είναι η απάντησή σας πάνω σε αυτό, διότι είσαστε εκτός, απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα τρίτο μέρος, πιο ουδέτερο. Ποιο είναι το, η άποψη σας για το μέλλον. Είπατε ότι η Καλιφόρνια δαπανά πάνω από αυτά που, από τα έσοδά της και επηρέασε την κατάσταση πολύ κρίση. Και βλέπουμε και την κατάσταση τη Ευρώπη. Οι νόμοι τη Ευρώπη διαφέρουν πολύ από τη ΣΥΠΑ. Είναι ομοσπονδιακή χώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το Τέξα είναι σε καλύτερη κατάσταση σαν πολιτεία. Και ίσω ε, το Τέξα θα μπορούσε να αγοράσει τίτλου τη Καλιφόρνια. Τι γίνεται λοιπόν ε, με το θέμα των ομολόγων με τους τόκους. Θα πρέπει να παραμείνει ένα όριο το 100% όπως έγινε και στην Ιρλανδία για το Senior Bond Interest. Το χρέος της Ιρλανδίας αυξήθηκε σημαντικά και αυτό πρέπει να βρεθεί μια λύση να διατηρείται το κεφάλαιο, να δημιουργείται κεφάλαιο μέσω νέων ομολόγων. Όταν Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές κατηγορίες χωρών. Υπάρχουν χώρες που εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας, με ίσως μείωση του ΑΕΠ τους επί σειρά ετών, με υψηλά επίπεδα ενεργείας και μετά θα είχαμε ένα άλλο στατόπεδο χωρών στην Ευρώπη, όπου θα σημειώνεται σημαντική ανάπτυξη, όπου τα επίπεδα απασχόλησης θα είναι καλά και μεγάλο ποσοστό θα υπάρχει και μεγάλο ποσό, ε, μεγάλος αριθμός εκρών από τις φτωχότερες των προ χώρες προς τις πλουσιότερες χώρες για να βρουν δουλειά. Ποια είναι η άποψή σας. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σενάριο όπως αυτό περιέγραψα στην Ευρώπη Μήπω φτάσουμε σε αυτό το στάδιο εδώ σε 10 χρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είχαμε μακροπρόθεσμη πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που ήθελε να καλύψει τα κενά μεταξύ των κρατών μελών. Αν εφαρμόσουμε λάθος μέτρα θα φτάσουμε στην κατάσταση που περιέγραψα. Ε, Πώ τα βλέπετε εσείς από τη σκοπιά των Ηνωμένων Πολιτειών την κατάσταση στην Ευρώπη. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα ερώτημα που να σας πω ειλικρινά δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμος ή σε θέση να απαντήσω. Αν ε, τα πούμε διμερώς μετά, αν μου δώσετε την κάρτα σας, ίσως θα μπορούσα να τα σκεφτώ αυτά που μου είπατε. Δεν είναι ο τομέας των γνώσεών μου, δεν νομίζω ότι έχω τις γνώσεις για να σας δώσω μια καλή απάντηση. Όσον αφορά την Καλιφόρνια, τα ομόλογα της Καλιφόρνιας, Μπορώ να σας πω ότι μπορούν να χρεοκοπήσουν πολιτείες της ΕΠΑ. Ε, στο τέλος τα senior bonds θα πληρωθούν με τους τόκους τους. Από ποιον ρωτάει ο πρόεδρος. Απάντησε. Οι δημόσιοι φορείς πληρώνονται ας πούμε μετά τις εκπαιδευτικές δαπάνες και λοιπά ο δημόσιος τομέας η υγεία, η περίθαλψη, τοπική αυτοδιοίκηση θα υποφέρουν οι άλλοι για να βγουν τα χρήματα για την εξόφληση του χρέους. Είναι η απάντηση. Νίκο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αγγελίδη, εγώ μιλάω πάντα ελληνικά. Υπογραμμίζω τη χαρά μου που είστε εδώ μαζί μας και την ελληνική σας καταγωγή για να πω ότι είναι ένας από τους λόγους που βρίσκω το κουράγιο να σας κάνω τις ερωτήσεις που θα σας κάνω. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι διέκρινα από την προφορική σας παρουσίαση ότι η Επιτροπή που δούλεψε υπό την Προεδρία σας έκανε μια έντιμη δουλειά και μάλιστα ορισμένα από τα συμπεράσματα με ευνηδιάσαν θετικά. Ερώτηση πρώτη λοιπόν. Διαπιστώσατε ότι η κρίση δεν ήταν αναπόφευκτη. Ρωτώ. Καλά. Δεν περίμενα να μελετούν στις Ηνωμένε Πολιτείε τον Μάρξ. Δεν ξέρω, το Χάρβαρτ και τα λοιπά, οι οικονομολόγοι, μάλλον τον είχατε αφήσει στην άκρη, τον ξεσκονίσαμε μετά την κρίση, έγινε best seller αλλού. Εντάξει. Τα σημάδια της κρίσης αυτού του μοντέλου, δηλαδή τη φούσκα των νέων τεχνολογιών, την κρίση στις τίγρης της Άπου δεν χτυπούσαν καμπανάκια ότι αυτό το σύστημα δεν είναι άμυρο, δεν είναι απαλλαγμένο από κρίσεις. Τόσος ήταν λοιπόν ο ιδεολογικός δογματισμός ότι αυτό το μοντέλο δεν θα έχει κρίσεις ή αν έχει θα είναι μικρές και διαχειρίσιμες. Και το ρωτώ όχι για την ιστορία. Όχι για την ιστορία εντάξει. Αλλά βγήκαν συμπεράσματα. Δηλαδή αυτό το βασικό δόγμα με το οποίο κινούνταν οι υπεύθυνοι, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Δηλαδή οι αγορές αυτορυθμίζονται. Ο ίδιος, από όσο ξέρω, έχω ακούσει, είπε μέα κούλπα. Ε, λάθος. Ναι, βγήκε το συμπέρασμα λοιπόν ότι δεν αυτορυθμίζονται οι αγορές και πρέπει να πάμε να δούμε άλλα μοντέλα. Δεύτερη ερώτηση που έχει σχέση με την ειλικρίνεια και την εντιμότητα των απαντήσεων. Ε, δεν είναι αστυνομικού χαρακτήρα. Με ποια κριτήρια φτιάχτηκε η Επιτροπή σας. Εμένα με εξέπληξε θετικά. Θα περίμενα και άλλα, αλλά αυτό είναι δικό. Εμεί, όπω ξέρετε και σα έχει ενημερώσει ο πρόεδρο, είμαστε κοινοβουλευτικοί. Εσεί με ποια κριτήρια φτιάχτηκε αυτή η επιτροπή που τόλμησε να πει ορισμένα πράγματα, άλλο αν δεν τηρούνται και ούτω κάθεξή. Τρίτη ερώτηση γρήγορα. Αυτή η υπεύθυνη, ο, ο, ο πρόεδρο των Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η οίκη αξιολόγηση. Εσεί δεν είχατε τη δυνατότητα. Τι θα γίνει με αυτού. Τιμωρήθηκαν. Είπατε, είσαστε κι εσεί απεσιόδοξο. Και η τελευταία ερώτηση, και δεν σα κουράζω. Πολλέ από τι τράπεζε των ηνωμένων πολιτειών δεν κατάλαβα ποιες και γιατί κάποιες σώθηκαν και κάποιες αφέθηκαν να καταρρεύσουν αλλά αυτό είναι ένα θέμα αμερικάνικο ουσιαστικά σώθηκαν με γενναίο δημόσιο χρήμα. Κατά μία έννοια κρατικοποιήθηκαν. Γιατί έπρεπε να ξαναγυρίσουν, αν είναι σωστή η πληροφόρησή μου, στους ιδιώτες που τη βούλιαξαν. Και εδώ δογματισμό. Ευχαριστώ ε, θα είχα και άλλες ερωτήσεις, αλλά εκτιμώ ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Uh, ευχαριστώ. Uh, first of all, the, um... Εγώ ευχαριστώ. In a sense, it lulled people... Υπήρχαν δείγματα του κινδύνου που οδήγησαν βέβαια τον κόσμο στο να πιστέψουν ότι η Federal Reserve μπορούσε να συγκρατήσει τη φούσκα. Και λέγανε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές είναι λιγότερο μετάβολες, πιο σταθερές και ότι δεν θα γινότανε αυτό το οποίο έγινε. Ναι, ναι, έξι-τρεις ήταν οι ζημιές. Και είχαμε αυτή την ύφεση που κράτησε σχετικά λίγο ένα χρόνο. Ούτε είχαμε τόσο τρομερές επιπτώσεις όσον αφορά την απασχόληση. Ούτε ήταν οι έμεσες συνέπειες τόσο μεγάλες, αλλά κοιτάξτε τι έγινε εκείνη την περίοδο. Είχαμε αυτές τις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από τις τράπεζες όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια που παρομοιάζουν ακριβώς με τα όσα έγιναν με αυτήν την φούσκα. Είχαμε κάποιες ε, εκθέσεις που τα λέγανε όλα Ρόδινα είχαμε κάποια σκάνδαλα είχαμε τράπεζες που πληρώσαν δις για να βοηθήσουν κάποιες εταιρείες σαν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους χωρίς να υπάρχει ενός είδους ε, ε, ανοιχτή διαδικασία όπως θα περίμενε κανείς. Επομένως, το 2001 2002-2003 είχαμε αυτό το κύμα των σκανδάλων. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα συναγερμός για το τι ερχόταν. Και είδαμε ότι χάσανε το πιο σπουδαίο οι Αμερικανοί, τα σπίτια τους. Και είχαμε έναν γερουσιαστή του Μέλλον που προσπάθησε κάτι να κάνει μετά από το σκάνδαλο τη Ένρων. Το Σαρμπάνι. Το Σαρμπάνι, οπότε να, ε, είμαστε και εθνικά περήφανοι σε σχέση με αυτό. Επομένω, ναι, υπήρχαν κάποιοι πρόδρομοι, πρόδρομα δείγματα τη κρίση. Κύριε Κλίντς είπε ότι θα προτείνω να σα το έχω πει. Να σα το πω τώρα. Ότι πρόκειται για μια επιτροπή με 10 μέλη και τελικά. Δεν ψηφίσαμε και οι 10, ναι, στην έκθεση. Οι 6 προέρχονται από τους ε, Δημοκράτες, 4 από τους Ρεπουμπλικάνους, τους όρισαν δηλαδή Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκράτες. Ήταν άτομα με εμπειρία ε, από τραπεζικές αλλαγές, από το κλάδο των στεγαστικών δανείων κλπ. Και τελικά οι δημοκράτες όρισαν πέντε δικούς τους και έναν εξάρτητο. Οι ρεπουμπλικάνοι τέσσερις δικούς τους και όταν ολοκληρώθηκε η έκθεση την προσυπέραψαν πέντε δημοκράτες και ένας ανεξάρτητος αλλά όμως οι ρεπουμπλικανοί δεν συνεφώνησαν. Ήταν διχασμένοι. γιατί θέλω να κατηγορηθεί η κυβέρνηση και επομένω ε, αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν συμφωνούσαν οι υπόλοιποι. Οι άλλοι τρει ε, ρεπουμπλικάνοι είπαν ότι συμφωνούσαν και έλεγαν ότι συμφωνούν όσοι επιτοπλίστων με αυτά που είπε η πλειοψηφία αλλά μεγαλύτερη διαφοροποίησή τους ήταν ότι συμφώνησαν όσον αφορά τις τράπεζες, συμφώνησαν για τα στεγαστικά, συμφώνησαν ότι υπήρχε δαπάνη, ε, υπήρχαν απάτες σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, όμως δεν συμφώνησαν για το ποιο είχε την ευθύνη που θεωρήσαμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας. Δεν ήταν απλώς να πούμε το τι έγινε, να πούμε για το γιατί συνέβη. Και τελικά ποιο είναι υπεύθυνος. Φυσικά και επιδεινώθηκαν τα στεγαστικά και τελικά ήταν επικίνδυνο το πώ γινόταν, γιατί είχαμε εκατομμύρια τέτοιων δανείων, τα οποία ευθύ εξ αρχή ήταν ελαττωματικά. Οπότε αρνήθηκαν την κατανομή των ευθυνών. Ε, ενώ εμεί του λέγαμε ότι η Κεντρική Τράπεζα μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε και αποφάσισε κακώ να μην κάνει τίποτα μέχρι τον Ιούλιο του 2008, τότε που έσκασε η φούσκα και πια είχαμε βυθιστεί στην κρίση. Άλλοι σώθηκαν, άλλοι όχι. Πρώτα πρώτα. Μικρότερες τράπεζες, επενδυτικές, η FDIC, σώθηκαν, εξαγοράστηκαν και από πιο σημαντικές δύο κατέρευσαν. Οι Lehman Brothers και η Washington Mutual. Δεύτερη περίπτωση κατά την οποία δεν ικανοποιήθηκαν οι πιστωτές. Η δε κυβέρνηση ποτέ δεν είχε ολοκληρωμένο σχέδιο. Περιπτωσιολογικά ενεργούσαν. Με την JP Morgan κατά περιπτώσεις ε, ε, βοηθήθηκαν ναι παντού χρωστάγανε και τελικά αφέθηκε η Λίμαν να καταρρεύσει όπως τα εξηγούμε στην έκθεση θεωρούμε ότι αφέθηκε να καταρρεύσει γιατί ο Μπερνάγκη ακόμα και σήμερα λέει και τον ε, εκτιμώ ότι δεν μπορούσαν να τους δανείσουν. Δεν είχαν αρκετή περιουσία ελέμαρ για να, για να δανείσουν χρήματα. Εγώ ότι είναι συνδυασμό πολιτικών αιτιών ε, μετά πως έγιναν με την ΜΕΙ, ΜΑΚ και σε συνδυασμό με το ότι δεν είχαν αρκετά ενετικά στοιχεία. Και τελικά θεώρησε ότι η αγορά θα εξισορροπηθεί από μόνη της αφού καταρρεύσει λίμα. Όχι, δεν υπήρχε κάποιο συνεχτικό σχέδιο. Με κάθε περίπτωση στο γόνατο την, την αντιμετώπιζαν. Και με την AIG πάλι το, το πρόβλημα ήταν το ίδιο. Οπότε ήταν συνειδητή η απόφαση της να μην σώσουν τη Λέμαν για όλους αυτούς τους λόγους. Ε, ίσως έχει αυτό επιρροή και στην ε, Goldman. Όχι, δεν νομίζω ότι κάποιος θα έπαιρνε μία απόφαση που θα είχε βλαπτικό αποτέλεσμα. Ε, τώρα εάν προχώρησαν βαθιά στα ε, παγωμένα νερά δεν είμαι σίγουρος αλλά ε, υπήρχαν ορισμένες αποφάσεις πολιτικές οι οποίες ήταν αμφιλεγόμενες σχετικά με τις διασώσεις. Το λόγο έχει τώρα ο Μάριο Μποργέζιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω την εκτίμησή μου για την παρουσία του εδώ, του Προέδρου του κ. Αγγελίδη. Τον ευχαριστώ και όπως και οι άλλοι. Και για την ιστορική σημασία που έχει συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας. Αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, η βασίλισσα της Βρετανίας σε μια σημαντική συνάντηση με την επιστημονική κοινότητα των Βρετανών οικονομολόγων έκανε ένα εκπληκτικό ερώτημα και του το έστειλε. Πώ κανεί από εσά δεν χτύπησε συνεγερμό, δεν έδωσε κάποιε ενδείξει, δεν προέβλεψε αυτό τον κατακλυσμό, τον οικονομικό που μα έπληξε. Αυτό ρώτησε η Βασίλισσα. Εμεί στην Επιτροπή μα, και εγώ το υπογράμμισα αυτό, υπενθυμίσαμε ότι το βραβείο Νόμπελ της οικονομίας της Γαλλικής ο Μωρίς Σαλέ είχε προβλέψει τα αίτια ο Γάλλος νομπελίστας, ε, είχε προβλέψει τα αίτια. Εγώ θέλω να ρωτήσω στην Επιτροπή σας τη είπα, διεφάνισαν κάποια στοιχεία επιστημονικά. Κάποιοι οικονομολόγοι που δεν εκτιμούσαν το σύστημα της Wall Street και τα διάφορα λόμπι, τέτοιοι οικονομολόγοι ε, το έθεσαν το θέμα. Και αναφέρομαι στις έντονες δράσεις στο λόμπι, γιατί Αληθεύει μεν αυτό που αναφέρει η έκθεσή σας ότι υπάρχει σκιώδε τραπεζικό σύστημα. Το 2008 ξεπέρασε το κανονικό σύστημα. Αυτό συνέβη κάτι στην κατάργηση των προστασιών και του τείχους που υπήρχε κατά τη, του, της ελευθερίας της κερδοσκοπίας εις βάρος των αποταμιευτών που προβλέπει ε, ο νόμος Κλάς Στίκαλ. Ερώτημά μου, η Επιτροπή σας δεν βλέπει να υπάρχει ανάγκη να επαναγκαθιδρυθεί, να επανατοποθετηθούν προδιαγραφές, νόμοι βάσει του νόμου Glass-Steagall διότι φάνηκε ότι οι διάφοροι λομπίστες συνδεόταν με την χρηματοστατική κερδοσκοπία και θέλαν να καταργηθεί αυτός ο νόμος. και οι διαμαρτυρίες που ακούγονται στην Ευρώπη είναι ε, αδύναμες. Λένε ότι αυτός ο νόμος θα ήταν καλά της ε, ε, παράδοσης των τραπεζών. Μέχρι την κατάρριξη του νόμου οι διατάξεις λειτουργούσαν μια χαρά. Δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι κάπως παράξενο αυτή η υπερχρηματοδότηση της, της ΦΕΔ ε, που χορηγείται αυτή η σούπερ χρηματοδότηση προς κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την τεράστια χρηματοδότηση. So, uh, let me take each of these. First of all... Απάντηση, να απαντήσω σε μία-μία ερωτήσει. Μιλήσαμε με διάφορους πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς. Κατά τις 740 περίπου συνεντεύξεις ε, ακούστηκαν ε, διάφοροι ακαδημαϊκοί, πολλοί προειδοποιούσαν για τις δυνατότητες κατάρρευσης του συστήματος. Στη σελίδα 17 της εκθέσεώς μας το βλέπετε αυτό αναφέρουμε εκεί ότι κάποιος με τους, ο... τους οποίους παραθέσαμε μάλλον ήταν ο Ρόγκαραμ Ρατζάν που πήσε στην ετήσια διάσκεψη της Federal Reserve στο Jackson Lake Lodge το 2005 και παρουσίασε ένα έγγραφο το 2005 με τίτλο «Η χρηματοπιστική ανάπτυξη έκανε πιο επικίνδυνο τον κόσμο». Είπατε ότι τα στελέχη από, ε, προσελκύονταν από βραχυπόδοσμα κέρδη και είπε ότι τα, κέρδη, τα, τα, κέρδη, τα credit swaps θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν το σύστημα και τα εθνιστικοί φορεί να ήταν αδύνατοι να, να διορθώσουν. Και υπενθύμησε στην FICC, που είναι η Επιτροπή Έρευνα για τι οικονομικέ κρίσει και είπε ότι ο υπουργό Οικονομικών δεσμένο, που ήταν πρόεδρο του Harvard University ε, είπε ότι ήταν αντίθετο στην τεχνολογική αλλαγή και έλεγε ότι αισθανόμουν σαν ένα Χριστιανό που είχε μπει σε, σε ένα συνέδριο ε, πεινασμένων λεόντων. Ε, και κάποιοι άλλοι ακαδημαϊκοί έγραψαν τότε και αναφέρθηκαν για την, στην επικείμενη κρίση οπότε είναι το ένα, υπαριθμόν ένα θέλετε στοιχείο ερώτημα 1. 2. Glass-Steagall, έτσι. Ρωτήσατε για τον νόμο Glass-Steagall. Ναι. Να πω το εξή. Ο τείχο αυτό αυτός Glass-Steagall άρχισε να καταραίει πριν γίνει η ανάκληση του νόμου το 1999. Τη δεκαετία του 1980 άρχισε να μην εφαρμόζεται από τη Federal Reserve επί Alan Greenspan. Οι τράπεζε μπορούσαν να κάνουν όλο και περισσότερο για όσον αφορά το εμπόριο αξιογράφων. Δεν μπορώ να πω γενική δήλωση, να πω κάτι γενικό πάνω σε αυτό. Να ένα παράδειγμα, να αμφισβήτητα, αν δείτε αυτά που συνέβησαν στη City Group, το παραδοσιακό αυτό τραπεζικό ίδρυμα, όπως έπεφταν η τύχη του Glass Steagall, ενεργοποιήθηκε πολύ στον τομέα των αξιογράφων, των securities, και αυτή ήταν η βασική πηγή των απολειών της περίπου 50 δις ευρώ. Όταν έφυγε ο τείχος, κινδύνευσε όλο το, το χρηματιστικό ίδρυμα. Δεν λέω ότι ήταν το αίτιο. Αλλά όσον αφορά την Citigroup, όταν έπεσε ο τείχο, η Citigroup ανέλαβε πολύ περισσότερου κινδύνου από ό,τι θα μπορούσε να κάνει αν υπήρχε ακόμα ο τείχο. Θυμηθείτε το Glass-Steagall. Ε, είναι σημαντικό στοιχείο. Όταν εφαρμόστηκε τη δεκαετία του 20, αφορούσε την προστασία των καταναλωτών. Είχε σχεδιαστεί για να προστατεύει του καταναλωτέ να μην πηγαίνουν σε μια τράπεζα που θεωρούσαν ότι ήταν συντηρητικό χρηματοστατικό ίδρυμα και τη δεκαετία του 20 να προσφέρει ομόλογα άκρος Για προστασία των καταναλωτών είχε θεσπιστεί ο νόμος, που είχαν, θεωρούσαν ότι αν πάει στην τράπεζα οι καταναλωτές αγόραζαν συντηρητικούς τίτλους. Ε, τρίτο ερώτημα, δεν θυμάμαι το τρίτο ερώτημα, το σημείωσα. Ποιο ήταν το τρίτο ερώτημα. Το κάλυψα, σας κάλυψα. Ωραία. Uh, το τρίτο ερώτημα. Το επαναλαμβάνετε το τρίτο ερώτημα. Εκτός μικροφώνου. το Τρίτο ερώτημα ήταν πώς η Fed επένδυσε, έδωσε τεράστιες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτό ήταν το ερώτημα. Απάντηση. Ρωτήστε τον κύριο Μπαρνέκη. Μπορέσαμε να δούμε πολλά από τα αρχεία των δανείων που έδωσαν στα χρηματιστικά ιδρύματα. Σας το πω ομά, μία από τις αντιρρήσεις μας, και ο κ. Σκρίντ θα, θα, θα συμφωνεί με αυτό, είχαμε πολύ λίγο χρόνο. Ιούλιο του 2009 μας έβαλα να ξεκινήσουμε. Έπρεπε να δημιουργήσουμε από το μηδέν ερευνητική ομάδα και έπρεπε να ετοιμάσουμε Δεκέμβριο του 2010 αρχικά έκθεση και Ιανουάριο 2011. Ανοίξαν πολλές πόρτες, ε, όπως είπα στις παρατηρήσεις μου ανοίξαμε πολλέ πόρτε. Τι εννοώ, εκθέσαμε πολλέ πληροφορίε που ήταν άγνωσε πριν. Όπω είπα στην αρχή, εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό, ανοίξαμε πολλέ πόρτε και η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί. Η Fed πρόσφατα, όπω γνωρίζετε, δημοσιοποίησε πολλά περισσότερα, πολλέ περισσότερε πληροφορίε για το ποιο χρησιμοποίησε τι δυνατότητε εκτόσεων και μειώσεων και χρειάζεται να δοθεί συνέχεια. Αν όχι από το Κογκρέσο, από κάποιο άλλο ερευνητικό φορέα ή ερευνητικού ε, φορεί. Ευχαριστώ. Και τώρα η ε, εκ νέου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, πολλά διδακτικά στοιχεία υπήρχαν σε αυτά που μας είπατε και επανέρχομαι στην εισαγωγή σας διότι ε, για αυτούς που μας ακούν, αυτούς που περιμένουν Υπάρχει ένα μήνυμα ότι θα αλλάξουν τα πράγματα ε, αλλά πολλοί ανησυχούν και φαντάζομαι ότι ε, αν τέλειωσε η δουλειά της δικιάς σας επιτροπής και η δικιά μας ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι το αποτέλεσμα αυτών των σχολείων είναι ότι οι πολιτικοί πρέπει να αντισταθούν στις αγορές και να μπορέσουν να επιβάλλουν στους παίκτες της αγοράς τα μέσα που χρειάζονται κατά τρόπον ώστε οι αγορές να λειτουργούν εύρυθμα. Και αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε σε εσά ε, και στα σχόλιά σας μας δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουμε στη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά το πακέτο της νομοθεσίας Φρανκ το οποίο έχει αποδυναμωθεί από το Κογκρέσο και που δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία σας καθησυχάζω. Τα ίδια περνάμε και εμείς, διότι για σας το πακέτο Dodd Frank υποσχόταν πολλά στη ρύθμιση. Εμείς έχουμε ένα πακέτο για την εποπτεία πολλά υποσχόμενο ε, και στην ρύθμιση. Αλλά για την εποπτεία αντιμετωπίσαμε τις ίδιες δυσκολίες με εσάς δηλαδή τα κράτη-μέλη άπαξ και δεχθήκανε ε, τον οργανισμό διεπίστωσαν ότι ε, τα πράγματα άλλαξαν όταν ε, χρειάστηκε να επιλογούν, επιλεγούν άτομα που έπρεπε να ε, έχουν μεν κύρος αλλά όχι υπερβολικό για να συμμετάσχουν στην εποπτεία. Απαντήσατε στη, στον συνάδελφο Μπογκέζη όσον αφορά το διαχωρισμό μεταξύ επενδυτικής τράπεζας και τράπεζης καταθέσεων και εγώ προβαίνω σε αυτό το διαχωρισμό στην τελική έκθεση και πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα πολύ προσεκτικά. Επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα πριν, τη συνέντευξη τύπου που οργανώσαμε Δηλαδή, όταν στην Επιτροπή αυτή ε, κρίσεως, στην ε, πρώτη προσωρινή μας έκθεση, είχα μία ολιστική ε, προσέγγιση όσον αφορά τις αιτίες της κρίσεως, μιλάμε για οικονομική, ε, χρηματική και κοινωνική κρίση, δηλαδή ουσιαστικά τα ίδια που περάσατε κι εσείς. Η πρώτη έκδοση την οποία είχα προτείνει σαν ανάλυση της κρίσεως προσέκρουσε σε αυτούς οι οποίοι ε, δεν ε, ήθελαν να αντιληφθούν τις κοινωνικές αιτίες της κρίσεως, δηλαδή ότι οι χρηματαγορές είχαν εκμεταλλευτεί τις πιέσεις στους μισθούς για να επιτρέψουν ε, την χρηματοδότηση και να δοθούν δάνεια σε άτομα με απίθανες και ανέφικτες συνθήκες και ε, όταν ε, ε, πρέπει κανείς να ελέγξει τις χρηματαγορές δεν υπάρχει συνένεση. Άρα η ιδέα ότι αυτοί που ευθύνονται για την κρίση θα πρέπει να βρουν και τη λύση δεν είναι εφικτή. Διότι όπως είπατε όλο το απόγευμα υπάρχει μία ρυθμιστική διαιτησία. Υπάρχει μία ισχύς των οργανωμένων λόμπι των χρηματαγορών και για να λειτουργήσει η δημοκρατία και οι αγορές μας πρέπει να οργανωθεί η αντίσταση και να επανέλθουμε στην ουσία της δημοκρατίας, δηλαδή να ε, επιτρέψουμε να υπάρξουν αντίβαρα. Και νομίζω ότι η έκθεσή σας ε, στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντική και ελπίζω ότι και εμείς θα συμβάλλουμε με την ε, εισαγωγή μας στο θέμα της κρίσεως. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος θα σας ευχαριστήσει ο ίδιος και αυτό συνάδει με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά μας δηλαδή μεθαύριο οι συνάδελφοι θα καταθέσουν τις τροπολογίες για την τελική έκθεση και άρα ε, οι εξηγήσει που μας δώσατε σήμερα το απόγευμα θα χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα από τους συναδέλφους και ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί ε, να αναταχθεί πλήρως η έκθεση ε, τουλάχιστον ε, αν κατάλαβα καλά το πνεύμα βάσει του οποίου μιλήσατε. Έχετε ακόμη φίλ τα ε, ακουστικά οπότε μπορώ να σας πω λίγα λόγια στη γλώσσα μου. Η Περβόνς πολύ σωστά σας είπε ότι κρατήσατε το λόγο σας. Στη Washington μας είχατε πει ότι θα έρθετε να μας επισκεφτείτε να μας παρουσιάσετε το αποτέλεσμα της εργασίας σας ε, το πράξατε. Είχαμε μια πολύ ανοιχτή συζήτηση. Μας εντυπωσίασε όχι μόνο ε, το αποτέλεσμα αλλά πόσο ανοιχτά και ειλικρινά ε, μας παρουσιάσατε πόσο καταλήξατε σε αυτό το αποτέλεσμα και αντιλαμβανόμαστε ότι σε πολλά θέματα έχουμε τις ίδιες απόψεις. Όχι μόνο όσον αφορά τις αιτίες της κρίσης υπερβών έθιξε τα θέματα αυτά αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τις ε, κοινωνικές δομές, τις κοινωνικές ανισότητες και είμαστε πεπισμένοι ότι όπως και εσείς ότι δεν έχει τελειώσει η κρίση και ότι χρειάζονται ε, πολιτιστικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν και ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπη Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε μία τόσο στενή συνεργασία μεταξύ όλων των μελών του G20 αλλά νομίζω ότι μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών μπορούμε να συνεργαστούμε κατά τρόπον ώστε ε, να αποφύγουμε ε, τους πειρασμούς που δημιουργεί αυτό το, αυτή η ρυθμιστική ε, διαιτησία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι αύριο πρέπει να να φύγετε για να συνεχίσετε την έρευνά σας και σε ευχόμαστε κάθε καλό αποτέλεσμα. Εγώ σας ευχαριστώ και πρέπει να σας πω ότι ήταν μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό προτέρημα για μένα να μπορέσω να έρθω εδώ, να σας μιλήσω και ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας είμαι χρήσιμος στη σκέψη σας και τέλος ελπίζουμε ε, όλοι ότι δεν θα, χρειαστεί δεν θα χρειαστεί να ξανασυγκληθούν αυτές οι επιτροπές ε, στην Αμερική και στην Ευρώπη για να εξετάσουμε μία τόσο καταστρεπτική κρίση. Από πολλές πλευρές ε, το πιο ουσιαστικό στοιχείο στην έκθεσή μας ήταν να ε, καταγράψουμε τα γεγονότα, το τι συνέβη τα τελευταία 30 χρόνια και τα γεγονότα είναι πολύ σημαντικά διότι μπορεί τα χρηματιστήρια και οι υπεύθυνοι ε, να κατακρίνανε τις απόψεις μας αλλά δεν αμφισβήτησαν την ακρίβεια των διαπιστώσεών μας και ελπίζουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε μια καλύτερη έκβαση στο μέλλον και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ.